Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση που είχαμε. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο σημείο 5. Παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της πρότασης αναδιατύπωσης της, ε, της, ε, της οδηγίας την επιστροφή του 2008. Αυτό το σημείο το έχουμε χωρίσει σε δύο μέρη. Θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης, περίπου 15 λεπτά, και στη συνέχεια θα έχουμε μια παρουσίαση του σχεδίου, τελική εκδοχή της μελέτης αρρηκτύπου του Κοινοβουλίου 15 λεπτά και επ' αυτού εάν ε, κάποιοι συνάδελφοι τώρα φεύγουν και δεν ενδιαφέρονται για το θέμα παρακαλώ να φεύγουν ησύχω. θα περάσουμε στο πρώτο μέρος και θα δώσω το λόγο στον εισηγητή την κυρία Σατζεντίνη την εισηγήτρια θα μας παρουσιάσει λοιπόν το σχέδιο έκθεσης για την οδηγία επιστροφών είναι και αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας και γι' αυτό είναι εδώ. Ε, έχει το λόγο. Φαντάστηκα ότι θα ήταν εξαιρετική η ευκαιρία που έχω να είμαι εδώ πάνω και να σας παρουσιάσω αυτή την έκθεση. Δεν θα σας κουράσω γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικότερο να ακούσουμε τους ε, ερευνητές μας ε, που διεξήγαγαν αυτή τη μελέτη αντικτύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την οποία εμεί ζητήσαμε γιατί δεν μα δεν μας απέστειλε σχετική μελέτη αντικτύπου η Κομισιόν. Στη συνέχεια ζητήσαμε και λάβαμε ανάλυση από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, από τον Ευρωπαίο Πόπτη Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και την Frontex και νομίζω ότι Απ' έξω τα λέω, αλλά νομίζω ότι δεν κάνω λάθο και κάναμε πάρα πολλές ε, συναντήσεις σκιωδών ήδη για να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε αρκετές γνώσεις ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το φάκελο και για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε και νέες ε, τάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με διαφάνεια. Γι' αυτό τον σκοπό, άλλωστε, έχω ε, καταρτήσει και ένα κατάλογο με τους οργανισμούς στους οποίους έχουμε έρθει σε επαφή και με τους οποίους έχουμε μιλήσει. Επίσης έχω συντάξει ένα επεξηγηματικό σημείο μας, το οποίο εξηγώ για ποιο λόγο έκανα τις επιλογές που έκανα. Και μία από τις επιλογές αυτές είναι ε, η τροποποίηση αυτής της νομικής πράξης. Αν και θα μπορούσε κανείς να πει ότι θα μπορούσαμε απλά να το γνωρίσουμε και να ε, συνεχίσουμε για να κάνουμε αυτά που είπε η Κομισιόν το 2017 όταν και εξέδωσε κάποιες συστάσεις και να πούμε κράτη-μέλη σας παρακαλούμε ξεκινήστε να υλοποιείτε την, την ισχύουσα οδηγία για τις επιστροφές προτού αρχίσουμε να τροποποιούμε την ισχύουσα νομοθεσία. επειδή πολλά από τα προβλήματα, και συμφωνώ με αυτό, που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη δεν σχετίζονται με την απουσία νομοθεσίας, αλλά με την ε, απουσία εφαρμογής αυτής. Καθώς λοιπόν η Κομισιόν υπέβαλε την πρότασή της και το Συμβούλιο συνεχίζει να ασκεί πιέσεις, εγώ αποφάσισα να δράξω αυτή την ευκαιρία και να ε, συντάξω μια οδηγία για τις επιστροφές η οποία θα κινείται, κινείται πλήρως και σαφώς εντός των ορίων του διεθνούς δικαίου και η οποία θα μπορεί πραγματικά να τεθεί σε εφαρμογή με αποτελεσματικότητα χωρίς να δημιουργεί φρούδες ελπίδες. Και αυτό το λέω και στο επεξηγηματικό σημείωμα μου. Ε, για το σκοπό αυτό ε, επέλεξα κάποιες προτεραιότητες Επικεντρώνομαι στις ε, ε, εθελοντικές ε, αναχωρήσεις και επιστροφές. Φυσικά υπάρχουν και οι καταναγκαστικές τέτοιες, γιατί δεν μπορεί κανείς να βασίζεται πλήρως στον εθελοντικό χαρακτήρα των επιστροφών, δίνοντας, την, αφαιρώντας από τις αρχές το τελικό στάδιο, το οποίο είναι η αναγκαστική επιστροφή. Όμως η Κομισιόν στη δική της πρόταση βασίζεται στον καταναγκασμό, στις, στις αναγκαστικές επιστροφές, στην προσωποκράτηση κτλ. Ε, δεν υπήρχε καθόλου αναφορά στις εθελοντικές επιστροφές και αναχωρήσεις στην πρότασή της. Νομίζω ότι το βασικό ζήτημα σε σχέση με τις αναχωρήσεις δεν μας ε, αφορά εμάς ε, τόσο, αλλά την τρίτη χώρα, τις τρίτες χώρες οι οποίες θα πρέπει να επανυποδεχθούν τους πολίτες τους. Και δεν νομίζω ότι μπορούμε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο όταν επικεντρωνόμαστε στις ε, αναγκαστικές επιστροφές. Αν παρακολουθήσει κανεί τι διαπραγματεύσει που έγιναν μεταξύ Αφρικανική Ένωση και Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει προθυμία από κάποιε αφρικανικέ χώρε να επανυποδεχθούν πολίτε του, αλλά αυτό όταν οι πολίτε επιστρέφουν εθελοντικά. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε αποτελεσματικοί, πρέπει να δώσουμε την ιδέουσα σημασία και στι εθελοντικέ επιστροφέ. Δεύτερον, προσπάθησα να αυξήσω την αποτελεσματικότητα και βιασιμότητα τη διαδικασία επιστροφή προσφέρεται δηλαδή στον επιστροφόμενο όταν επιστρέφει στο, στην πατρίδα του. Μπορεί να επανενταχθεί στην κοινωνία του. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα επανενταχθεί στην κοινωνία του και δεν θα προσπαθήσει να ξαναγυρίσει με την πρώτη ευκαιρία. Γιατί αν έχει χρέη και ο μόνο τρόπο να τα αποπληρώσει είναι δουλεύοντα στην Ευρώπη, θα ξαναπροσπαθήσει να έρθει. Οπότε προσπαθήσαμε να αυξήσουμε αυτή τη βιωσιμότητα και την πρακτική εφαρμοσιμότητα. Έχει έγκυα σε σχέση με τι διαδικασίε επιστροφών. Α είμαστε ειλικρινεί. Όταν κανεί υποβάλλει αίτηση ασύλου, μπορεί να είναι και η δεύτερη φορά που το κάνει, αλλά πάντω βρίσκεται στη διαδικασία ακόμη, δεν μπορούμε να ζητούμε από αυτόν τον άνθρωπο να ξεκινά να ε, προετοιμάζει την επιστροφή του, να πάει δηλαδή στην προσβία του και να ζητήσει χαρτιά όταν ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί οριστικά ότι ε, απορρίπτεται ή εγκρίνεται η αίτηση ασύλου. Γιατί θέτουμε σε κίνδυνο ανθρώπου, όχι μόνο αυτού που ετούνται το άσυλο, αλλά και την οικογένειά του στην τρίτη χώρα. Μπορεί κάποιο να ήταν άγνωστο ότι είχε φύγει από τη χώρα ή να ήταν γνωστό αλλά χωρίς να ξέρουν, ότι έχει φύγει από τη χώρα του, αλλά χωρίς να ξέρουν οι αρχέ τη χώρα του που ακριβώ βρίσκεται. Να σα θυμίσω την υπόθεση ε, στην Κωνσταντινούπολη με τον ε, δημοσιογράφο από τη Σαουδική Αραβία που έχασε την ζωή του μέσα στην πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας. Αλλά δεν γίνεται να θέτουμε σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων. Επίσης, βάζουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια του παιδιού, εξασφαλίζοντας ότι τηρούνται όλες ε, οι πράξεις του διεθνούς δικαίου, νομικές, και ότι δεν θα προβλέπεται κράτηση παιδιών. Όταν υπάρχουν οικογένειες με παιδιά, δεν μπορούν αυτές να κρατούνται. Επίσης, προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε την αναλογικότητα, την συνεκτικότητα της νομοθεσίας και έκανα και κανένα δυο δραστικά πράγματα. Αφαίρεσα τη διαδικασία στα σύνορα. Και γιατί όσο δεν έχουμε σαφήνεια όσον αφορά την ε, διαδικασία στα σύνορα, στην νομοθεσία για το άσυλο, δεν μπορούμε να βάλουμε κάτι αντίστοιχο στην νομοθεσία για τις επιστροφές. Επίσης, άλλαξα τις απαιτήσει συνεργασίας στη διαδικασία για να ξεκαθαρίσουμε τι τελικά μπορεί κανείς να περιμένει όταν θα βρίσκεται στη φάση επιστροφής του, ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του, αλλά αφαίρεσα τις ε, περιτές απαιτήσει ε, και προϋποθέσεις για τη συνεργασία. Όλα αυτά λοιπόν κατέληξαν στη σύνταξη 120 τροπολογιών από την πλευρά μου. Νομίζω ότι ήμουν αρκετά διεξοδική στο έργο μου, αλλά βεβαίως ε, ευπρόσδεκτη κάθε πρόταση και από εσά. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 7η Φεβρουαρίου και ελπίζω να καταφέρετε να αξιοποιήσετε για τυχόν τροπολογίες και την μελέτη αντικτύπου που θα έχουμε την τιμή και την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σήμερα. Ευχαριστώ, Τζούντιθ. Περνάμε στους Κιώδης, Αναμαρία, για, εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως σκιώδης του ΕΛΚ χαιρετίζω αυτή την αναδιατύπωση της οδηγίας για τις επιστροφές που είναι απαραίτητη και εγώ ε, συνεργάστηκα για την μελέτη αντικτύπου. Χρειαζόμαστε μια πιο αποτελεσματική ενωσιακή πολιτική για την επιστροφή υπηκών τρίτων χωρών που δεν χρειάζονται διεθνή προστασία και γι' αυτό το λόγο δεν έχουν δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναδιατύπωση που προτείνει η Κομισιόν είναι μια καλή αφετηρία με θετικέ αλλαγέ. Για παράδειγμα, η ενίσχυση τη συνεργασία με τι χώρε προέλευση και την υποχρέωση των κρατών μελών να θεσπίζουν προγράμματα επιστροφών σε συνεργασία με τρίτες χώρες. Συμφωνώ, Τζούντιθ, μαζί σου ότι οι εθελοντικές επιστροφές θα πρέπει να είναι ο κύριος στόχος και θα πρέπει να εθαρρύνονται. Φυσικά πρόκειται για μακροπρόθεσμη λύση και αυτή είναι και καλύτερη. Όμως δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αποκλείσουμε και τις αναγκαστικές επιστροφές. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, θα υπάρξουν και τέτοιες και χαίρομαι που το είπες στην παρέμβασή σου. Ακόμη και για εκείνους για εκείνε όμω τι αναγκαστικέ επιστροφέ χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συνεργασία με τι χώρε καταγωγή, προέλευση, χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία με, μεταξύ των κρατών μελών μέσω τη ε, βάση δεδομένων διαλειτουργικότητα και χρειάζεται να παρακολουθούνται οι αποφάσει αλλά και οι δευτερογενεί μετακινήσει μεταξύ των κρατών μελών και να εξασφαλίζουμε ότι όλε αυτέ οι διαδικασίε θα εφαρμόζονται αποτελεσματικά. Ω ΕΛΚ, λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε αυτή τη διάσταση του θέματο και θα, θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτέ οι διατάξει δεν θα έχουν αρνητικέ επιπτώσει σε ευάλωτε ομάδε. Για παράδειγμα, θέλουμε να εντάξουμε μια καθαρή διάσταση φύλου στις διαδικασίες που δεν ε, λείπει τελείω από την πρόταση, αλλά να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες θύματα του τράφικινγκ και σεξουαλικής βίας. Όσον αφορά τα παιδιά, με χαρά βλέπω ότι η συγγήτρια έχει υιοθετήσει μια ε, προσέγγιση ε, για την αύξηση της προστασίας των παιδιών. Εμείς θα προτείνουμε την απαγόρευση κράτησης παιδιών και ε, να λαμβάνεται υπόψη ο ευάλωτος χαρακτήρας των παιδιών ο ευάλωτο χαρακτήρα δηλαδή να είναι το βασικό στοιχείο στη λήψη αποφάσεων. Τώρα, θέλω να επισέλθω σε κάποια συγκεκριμένα άρθρα, Όπω για παράδειγμα το άρθρο 6, της ε, επανεπιστροφής και της, ε, της ε, απαγωγής παιδιών. Καταλαβαίνουμε τις κινήσεις που έχει λάβει η Κομισιόν, αλλά ε, ο κατάλογος που έχει καταρτήσει δεν είναι επαρκής. Υπάρχουν για παράδειγμα ε, αναφορές στην παράνομη είσοδο, στην, στην ε, ε, απουσία ε, οικονομικών πόρων. Δεν είναι αντικειμενικά αυτά τα κριτήρια. Ωστόσο εμείς δεν δεχόμαστε, όπως προτείνει η συγκίτρια, να διαγραφεί πλήρως το άρθρο. Πρέπει να ε, ξεκαθαριστεί ότι αυτές οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κατά περίπτωση και κατά τόμου. για τον κίνδυνο διαφυγής. Όλα αυτά βεβαίω θα πρέπει να γίνουν με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ε, το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τη διαφυγή βεβαίω για να, για να καταπολεμηθεί ο, ο κίνδυνος διαφυγής δεν μπορούν να ξανακλείσουν τα σύνορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να εξαιρούνται τα παιδιά και να ε, παραπέμπονται στα εθνικά συστήματα προστασία του παιδιού. Και θα πρέπει ε, να απαγορεύεται για παιδιά ούτε καν ως έσχατο μέσο να χρησιμοποιούνται αυτά τα μέσα ενώ οι οικογένειε με παιδιά για την κράτηση θα πρέπει να, οι με παιδιά θα πρέπει να ε, φιλοξενούνται σε εναλλακτικέ δομέ. Άρθρο 9. Θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει δυνατότητα και για παιδιά, ακόμη και αν κάποιο υπήκοστη τη χώρα βρίσκεται σε κράτηση. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι σαφέ. Για την απαγόρευση εισόδου, το άρθρο 13, αυτό θα πρέπει να, ε, από αυτό θα πρέπει να εξαιρούνται τα παιδιά. Επίση, πρέπει να ενισχύσουμε το δικαίωμα πληροφόρηση των υπηκών τρίτων χωρών, που θα πρέπει να συμβαδίζει με τις εθελοντικές ε, επιστροφές. Και για τις επιπτώσεις άρνησης συνεργασίας, άρθρο 7, εδώ θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι τα δικαιώματά τους και οι υποχρεώσεις τους. Και τελευταίο, για τα παιδιά. Οι πληροφορίες που παρέχονται στα παιδιά θα πρέπει να είναι φιλικές προς τα παιδιά και σε γλώσσα και διατύπωση που μπορούν να κατανοήσουν οι δε επιπτώσεις μη συνεργασία δεν θα πρέπει, ε, δεν θα πρέπει μάλλον να υπάρχουν επιπτώσεις ε, σε παιδιά αρνητικές για τη μη συνεργασία τους αυτά. Ε, έχουν γίνει και πολλές συναντήσεις σκιωδών, συναντήσεις με πολλούς οργανισμούς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν πάρα πολύ χρήσιμες και ελπίζω συνάδελφοι να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε καλούς συμβασμούς σε κάποια βασικά ζητήματα, να προχωρήσουμε ε, γρήγορα και να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα έως το τέλος της θητείας. Ευχαριστούμε Αναμαρία. Να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Η Σιλβί Γιόμ δεν είναι εδώ, γι' αυτό και θα σας μιλήσω εκ μέρους της στα αγγλικά. Συνάδελφοι, η κυρία Γκυγιόμ θέλει να ζητήσει συγγνώμη, δεν μπορεί να βρίσκεται εδώ τώρα, λόγω ενεργημένων υποχρεώσεων στην εκλογική της περιφέρεια. Ως σκιώδης εισηγήτρια για την οδηγία περί επιστροφών από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες θέλει να ευχαριστήσει την εισηγήτρια. Η σύνταξη της έκθεσης προχωράει και η κυρία Γκυγιόμ εκτιμά πολλά από τα στοιχεία που έχει συμπεριλάβει η κυρία Σαρχεντίνη. Η κυρία Γκυγιόμ θα υποβάλει τροπολογίες συγκεκριμένα για το θέμα της επανένταξης, της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες και των συνοριακών διαδικασιών υποστηρίζει ότι καλό θα ήταν να έχουμε μια αποτελεσματικότερη πολιτική επιστροφών, όμω με προτεραιότητα τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραμεληθεί. Επίση, οι κρατήσει θα πρέπει να είναι λύση τελευταίου καταφυγίου, όπω λέμε, και να απαγορεύονται για την περίπτωση των παιδιών. Αυτά. Η ε, κυρία Γκυγιώμα ανυπομονή για να προχωρήσουν οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις. Ευχαριστούμε, κυρία Κάθμαν, Η κυρία Ίντβελτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Καλωσορίζουμε την πρόταση και τη γενικότερη κατεύθυνση που έχει ακολουθήσει η συγγήτρια. Θέλω όμως πολύ σύντομα να πω κάτι και για το πλαίσιο, το σκηνικό που εντάσσεται όλη αυτή η πρόταση. Διότι πραγματικά ε, ειλικρινώς το όλο σύστημα του ασύλου έχει κολλήσει στο Συμβούλιο τι εδώ και δύο χρόνια. Τίποτα δεν γίνεται. Τα θέματα που θέλαμε να επιλύσουμε με την πρόταση αναδιατύπωσης ε, ουσιαστικά στο πακέτο του ασύλου με τις δευτεραγιονείς μετακινήσεις ή τις περιπτώσεις υποδοχής που είχε κοιτάξει η κυρία Σίπελ είναι θέματα που θα μπορούσαν να επιληθούν εδώ. Είναι αλλαγέ που προτείνονται από την οδηγία των επιστροφών. Τελευταία στιγμή έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μίση Καρδιά και μας προτείνει αυτά ε, και λέει ότι δεν φταίμε εμεί που δεν έχει προχωρήσει το θέμα, αλλά τα κράτη-μέλη. Και όχι απλώς διαφωνώ μαζί τους ε, επί τη ουσία, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποτίθεται θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τα κράτη-μέλη. Οπότε Πραγματικά ελπίζω να εργαστούμε πολύ σοβαρά και επιμελώ. επί του ντοσιέ αυτού. Υποστηρίζω την όλη κατεύθυνση, τον προσανατολισμό τη εξηγήτρια και θα φροντίσουμε να υποβάλουμε σχετικέ τροπολογίες. Επιμένω όμω, δεν μπορούμε να ξεχνάμε εντελώ ότι το ντοσιέ αυτό σχετίζεται με τα υπόλοιπα ζητήματα που θα έπρεπε να βρίσκονται επιτάπητο. Αρνούμε να εργαστώ αποκλειστικώ για την εξωτερική διάσταση των πολιτικών ασύλου και μετανάστευση ενώ η εσωτερική διάσταση είναι εντελώς μπλοκαρισμένη λόγω της ε, ε, έλλειψης ε, ανάληψη ευθυνών από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Ευχαριστούμε, Σόφη. Η Επιτροπή θέλει πάλι το λόγο για να ολοκληρώσει, κύριε Ρότεμπεργκ. Θα μου πείτε αν θελήσετε να παρέμβετε. Κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την άριστη δουλειά της και όλος ιδιαιτέρως επειδή ήταν σχολαστικότατες και ευρύτατες οι διαπραγματεύσεις και οι συζητήσεις που είχαμε για να καταλήξουμε στη συνταξιματιφρά τους ε, εμπειρογνώμονες και όσου ε, προέρχονται από την κοινότητα των πολιτών για να μιλήσουν για τα θέματα αυτά. Με του κοιόδη εισηγητέ θα υποστηρίξω κάποιε τοπολογίε που έχει προτείνει και η εισηγητρία, κυρίω για την απάλληψη των κριτηρίων που καθορίζουν το ποιε περιπτώσει είναι περιπτώσει ε, διαφυγή. Θα δούμε ε, τα κράτη-μέλη πώ θα μπορέσουν να διοργανώσουν την εθελοντική και νόμιμη αναχώρηση και θα πρέπει να υπάρχει υπαρκή ε, συνοδεία καθ' όλη τη διαδικασία τη επιστροφή. Επίση, οι τροπολογίε θα πρέπει να ενισχύουν το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων που ε, λαμβάνουν απόφαση υποχρεωτικού επαναπατρισμού και μάλιστα αυτό να γίνεται αμέσω. Επίση, απάλληψη τη υποχρέωση συνεργασία των ε, της υποχρέωσης των, της συνεργασίας των πολιτών τρίτων χωρών, διότι μπορεί να αποκλειστούν από την συμμετοχή στα προγράμματα επανένταξης ε, που μπορεί να υπάρχουν. Επίσης, ε, περιορισμός στο ελάχιστο των ε, καταναγκαστικών επιστροφών και κατάρριξη των κρατήσεων. Επίσης, όχι κράτηση σε, μονο, σε κελιά, σε κλειστούς χώρους και περιορισμένους. Επίσης, πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, το εκπαιδευτικό σύστημα και κατάλληλη προστασία ανελίκων. Ταυτόχρονα, υιοθέτηση του της ε, υπεράσπισης κατά, κατά την παράθεση. Δηλαδή, οι πολίτε να μπορούν να παρουσιάζουν τα δικαιώματα της σε μια ακρόαση, την υπόθεσή του σε μια ακρόαση, σε περίπτωση που εξετάζεται η υπόθεσή του. Θα πρέπει το όλο δίκαιο να βασίζεται στο σεβασμό των θεμελιδών δικαιωμάτων. Πράγμα που μα επιφέρει την, ευθύ, την υποχρέωση να παρακολουθούμε όχι μόνο το σύστημα των υποχρεωτικών επιστροφών, αλλά και όλο το σύστημα του επαναπατρισμού. Δεν μπορεί αυτά να γίνονται επί τόπου χωρίς προειδοποίηση, ε, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια προσωρινή προετοιμασία έστω, ε, πρώτερη προετοιμασία, ε, διότι θα πρέπει όλοι οι πολίτες που πρόκειται να επιστραφούν να το γνωρίζουν, ακόμη και σε συνθήκες κράτησης. Θα πρέπει λοιπόν να λαμβάνουν γνώση και το Κοινοβούλιο και οι Εθνικέ Βουλέ. Επίση, κατάργηση του άρθρου 21 που δίνει το δικαίωμα στα κράτη-μέλη να ε, παρεκκλίνουν κάποιων διατάξεων της οδηγίας σε περιπτώσεις που υπάρχουν επίγουσες ανάγκες. Ε, περιπτώσεις ενοτεράς βίας, ε, όταν ε, μπορεί να κρατήσει περισσότερο καιρό η κράτηση α πούμε και τελικά να μην σέβονται την υποχρέωση που προβλέπει το άρθρο 19 στην παράγραφο 1 να χωρίζουν του μετανάστε από του ε, απλούς κρατουμένους και φυλακισμένου σε περίπτωση κράτηση σε σοφρονιστικά ιδρύματα. Ελπίζω αυτέ οι προτάσει μαζί και με τι υπόλοιπε από τι τροπολογίε μου και αυτέ τη ηγητρία να τύχουν τη απαραίτητη στήριξη ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε σε μια γρήγορη αναδιατύπωση τη οδηγία που να σέβεται τι ευθύνε και τι υποχρεώσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση από το Διεθνέ Δίκαιο σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Μπάρμπαρα. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε το γύρο των σκιωδών. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Εάν όχι, θα επιστρέψω στη Γιούντις, αλλά προηγουμένως ο κύριος Ρότεμπεκ από την Γενική Διεύθυνση Home. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να πάρω το λόγο. Θα παρουσιάσω σύντομα το σκεπτικό της πρότασης της Επιτροπής. Η πρόταση αυτή αναδιατύπωσης της οδηγίας για τις επιστροφές ξεκινάει από τη διαπίστωση ότι τα κράτη-μέλη έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά εμπόδια, πολλές δυσκολίες για να υλοποιήσουν μια πολιτική επιστροφών που να είναι αποτελεσματική Οπότε είναι απαραίτητο να προσπαθήσουμε να υπερβούμε αυτά τα εμπόδια και τους φραγμούς. Όλα αυτά βεβαίως με πλήρη σεβασμό των ε, θεμελιωδών αρχών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των αρχών της μη επαναπρόθεσης. Κατανοώ ότι το σχέδιο έκθεσης δεν ακολουθεί ακριβώς το ίδιο σκεπτικό, την ίδια συλλογιστική με την ε, δική μας την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζω όμως ότι με τις συζητήσεις που θα έχουμε, προσεχώς, θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε κάποιες παρανοήσεις που ίσως προέκυψαν. Ένα και μόνο παράδειγμα θα σας δώσω σε ό,τι αφορά την προτεραιότητα που θα δώσουμε στις οικειοθελείς επιστροφές. Ε, βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να γίνονται έτσι οι επιστροφές. Και όπως είπε και η συγγήτρια, οι οικειοθελείς επιστροφές θα αφορά τους ε, παράτυπους μετανάστες μόνο εφόσον απειλούνται από καταναγκαστική επιστροφή και απομάκρυνση. Η πρόταση της Επιτροπής δεν σημαίνει ότι όσοι έχουν ε, ταξινομηθεί ως κρατούμενοι δεν θα έχουν δικαίωμα πρόσβαση στο σύστημα των οικειοθελών αναχωρήσεων, οικειοθελών επιστροφών. Ο καθένα, οποιοδήποτε στάδιο τη διαδικασία, θα έχει πρόσβαση στο σύστημα των οικειοθελών επιστροφών. Αυτό επιδιώκουμε και μοχθούμε να πετύχουμε Στη φάση αυτή δεν θέλω να πω περισσότερα, απλώς θέλω να υπογραμμίσω αυτό το παράδειγμα. Μόνον σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ και να δω απλώς αν θέλει τίποτα να πει και η Προεδρία του Συμβουλίου. Όχι. Δεν χρειάζεται, αν δεν θέλετε. Ωραία. Γιούντιθ, θες πάλι το λόγο. Γιατί το είπα αυτό. Γιατί προσπαθούμε εδώ ως Κοινοβούλιο στη θητεία μας να προλάβουμε να πάμε σε διαπραγματεύσει με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμία μελέτη αντικτύπου για τίποτα, ε, οι πληροφορίε δεν είναι σαφεί. Τώρα λοιπόν, όταν ξεκινάει η διαδικασία, πώ μπορείτε να λέτε ότι παρανόμα αυτά που έχετε υποβάλει ω προτάσει. Εγώ πραγματικά δεν το δέχομαι αυτό. Υπάρχει χρόνο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για το Συμβούλιο, μόλι ε, το Κοινοβούλιο διαμορφώσει τη διαπραγματευτική του εντολή, να προχωρήσουμε. Εγώ εκτιμώ τι παρατηρήσει που έκαναν οι συνάδελφοι και ανυπομονώ για τι ε, τροπολογίε που θα λάβω. Θα κοιτάξουμε να τι διαμορφώσουμε σε συμβαστικέ λύσει. Μετά θα ψηφίσουμε και τότε θα έρθει στιγμή να μιλήσουμε με την Επιτροπή και το Συμβούλιο δούμε αν έχουμε διαφορετική προσέγγιση, αν ερμηνεύουμε τα πράγματα διαφορετικά και τότε θα κοιτάξουμε να έχουμε ένα κείμενο που να είναι καθαρό και τίμιο. Ε, κατά τα άλλα, δεν θέλω να επηρεάσω την όλη διαδικασία μα, ούτε θα δεχτώ τέτοιε εξωτερικέ επιδράσει. Ναι. Δεν βλέπω να λένε τίποτα τώρα όμω, έτσι κι το Συμβουλίο. Ωραία. Και τώρα να περάσουμε στο δεύτερο μέρο. Θε να πει κάτι άλλο για το κείμενο. Όχι, να περάσουμε λοιπόν στο δεύτερο κομμάτι, την παρουσίαση δηλαδή του σχεδίου τελικής εκδοχής της εστιασμένης της αντικτύπου του Ευρωκοινοβουλίου για την πρόταση για τις επιστροφές έγινε από κοινού από την Πανεπιστήμιο του Λόβεν, αυτό είναι το νομικό σκέλος, και το γραφείο Μιλιό που αφορά το οικονομικό σκέλος. Όλα αυτά υπό το συντονισμό ε, της μελέτης ε, ε, της μονάδας μελέτης, μελετών αντικτύπου εξ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του, της υπηρεσίας ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα δώσω αμέσως το λόγο στους ομιλητές για να παρουσιάσουν αυτό το, το τελικό σχέδιο μελέτης 15 λεπτά συνολικά παρακαλώ πρώτα η Καταρίνα, η Καταρίνα Άιζελε από την υπηρεσία ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχετε εδώ τη δυνατότητα να παρουσιάσετε και το PowerPoint. Σας παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ μα ζήτησε να δημιουργήσουμε μια μελέτη εκτύπου για την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλλον για την ε, αναδιατύπωση τη ε, οδηγία για τι επιστροφέ. Αυτή η πρόταση δεν συνοδεύτηκε από μελέτη αντικτύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπήρχαν και κάποια νομικά ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν και γι' αυτό ήρθαμε σε επαφή με την Ελίζ Μουίρ από την Πανεπιστήμιο του Λόβεν που είναι εμπειρογνώμονα σε συστήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων αλλά και οικονομικά ζητήματα για τα οποία ήρθαμε σε επαφή με την κυρία Μίνα Φερνάντες από την, το Γραφείο Εμπειρογνωμόνων Μιλιού σε ζητήματα ασύλου. Σύμφωνα με τη μελέτη αντικτύπου, το, το εγχειρίδιο της μελέτη αντικτύπου ε, του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή μας αποφάσισε το πεδίο που θα καλύψουν αυτή η μελέτη μαζί με τη μονάδα μελετών αντικτύπου εξάντε. Πρόκειται για μια εστιασμένη μελέτη αντικτύπου. Όπως ζητήθηκε από την Επιτροπή, οι πιο σημαντικές διατάξεις ε, της πρότασης της Κομισιόν αναλύθηκαν ε, σε σχέση με το status quo δεν εξετάστηκαν άλλε εναλλακτικέ, διότι ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που είχαμε στη διάθεσή μα. Μιλάμε εδώ για δύο μήνες, λίγο πολύ. Αυτή η εστιασμένη μελέτη αντικτύπου φτάνει στα, πέντε, στα εξής πέντε σημαντικά ευρήματα. Πρώτον, δεν, υπάρχει σαφή, δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία που να υποστηρίζουν την άποψη της Κομισιόν ότι η πρότασή της θα οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικές επιστροφές παράτυπων μεταναστών. Δεύτερον, η πρόταση πληρεί σε γενικές γραμμές την αρχή της επικουρικότητας, όμως κάποιες διατάξεις δημιουργούν ζητήματα αναλογικότητας. Τρίτον, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έχει έναν αντίκτυπο σε μια σειρά ανθρώπινο, ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων παράτυπων μεταναστών, μεταξύ των οποίων και ενδεχόμενη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τέταρτον, η πρόταση θα οδηγήσει σε ουσιαστικό κόστος και για τα κράτη-μέλη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα οδηγήσει δηλαδή σε έξοδα. Και πέμπτον και τελευταίο, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιουργεί ερωτηματικά σε ό,τι αφορά τη συνέπειά τη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές νομοθεσίες που εξετάζονται και εδώ, σε αυτή την Επιτροπή, όλες ιδιαίτερες εφόσον αυτή η ευρωπαϊκή νομοθεσία εκρεμεί. Θα δώσω τώρα το λόγο στην καθηγήτρια Μούιρ και στη συνέχεια την κυρία Φερνάντε και στη συνέχεια θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε και τα ερωτήματά σας. Um, um, Ευχαριστώ την κυρία Άιζελε. Ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μα δίνετε να παρουσιάσουμε τα συμπεράσματά μα ε, για το νομικό αντίκτυπο. Πρώτα για τη μεθοδολογία. Πρόκειται για εστιασμένη μελέτη αντικτύπου, οπότε ε, εξετάσαμε κάποια ζητήματα μόνο, εξετάσαμε τις διάφορες πηγές, ε, τι νομικέ που περιλαμβάνονται στη μελέτη αντικτύπου και σε επίπεδο μεθόδου εμείς πάντα ξεκινούμε από τον ορισμό των βασικών νομικών ε, όρων πριν εξετάσουμε τα τέσσερα ζητήματα αποτελεσματικότητα, αναλογικότητα, ε, επικουρικότητα και ανθρώπινα δικαιώματα και συνέπεια. Σε σχέση με το ερώτημα σας που μας, που μας θέσατε, αν δηλαδή αυτή η πρόταση δημιουργεί ε, ε πετυχαίνει το στόχο μια πιο αποτελεσματική επιστροφή. Το θέμα τη αποτελεσματικότητα είναι, είναι μια έννοια πολύ δύσκολη, πολύ λεπτή για τους ε, νομικούς. Εξετάσαμε λοιπόν τη συνέπεια της αφήγηση της Κομισιόν για το πώ προσεγγίζουμε την αποτελεσματικότητα τη πολιτική επιστροφών τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Η Κομισιόν λοιπόν έχει ορίσει στο μνημόνιο την αποτελεσματικότητα ω αύξηση του ποσοστού επιστροφών. Ε, έτσι λοιπόν πολλά είχαν ήδη, το είχαμε ήδη προκαταλάβει σε άλλα νομοθετήματα, αλλά μπορούμε να, εδώ να κάνουμε ένα σχόλιο. Αλλάζει εδώ ο τόνος, ε, είναι πολύ περιορισμένη η δυνατότητα εθελοντικής επιστροφής, αυτό είναι μια αλλαγή προσέγγιση της Κομισιόν, καθώς συνδέεται και με την επιλογή των κριτηρίων ε, για το κατάλογο, το, το κίνδυνο εξαφάνισης, αδιαφυγής τέλο πάντων, καθώς και ένα νέο λογοκράτησης όταν υπάρχει κίνδυνος για την δημόσια ασφάλεια και την εθνική ασφάλεια. Ε, το άλλο που μας ζητήσει να εξετάσουμε είναι κατά πόσο η πρόταση της Κομισιόν ε, σέβεται την αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Η πρόταση συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας και στο σύνολό τη και με την αρχή της αναλογικότητας. Όμως έχουμε ε, δει ότι υπάρχουν κάποιες, διατάξει διατάξεις που δημιουργούν ανησυχίες σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση με την αναλογικότητα. Και μπορείτε να τα δείτε εδώ μπροστά σα. Η απαγόρευση να υπάρχει μια περίοδο εθελοντικής ε, αναχώρηση, ο περιορισμό τη προσφυγή σε ένα μόνο επίπεδο, ε, πολύ περιορισμένο χρονικό ορίζοντα ορίζοντας για τι προσφυγέ και ε, βεβαίω η έλλειψη δεδομένων. Το γεγονό ότι δεν έχουμε αρκετά δεδομένα για να γίνει μια σαφή αξιολόγηση τη αναλογικότητα των μέτρων. Σε ό,τι αφορά το τρίτο σημείο τώρα, τον αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα και στα κοινωνικά, κοινωνικά δικαιώματα σε ό,τι αφορά αυτή την πρόταση. Για άλλη μια φορά έπρεπε εδώ να κάνουμε μια επιλογή ποια θεμελιώδη δικαιώματα θα εξετάσουμε, όπω άλλωστε συμφωνήθηκε και στην Επιτροπή. Ε, μια σειρά από θεμελιώδη δικαιώματα θα μπορούσαν να επηρεαστούν από συγκεκριμένε διατάξει όπω έχουν αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά τη διατάξει για την κράτηση, σίγουρα θα αυξήσουν τον κίνδυνο ε, μεροληπτικών ε, κρατήσεων Επίσης, η υποχρέωση συνεργασίας, όπως έχει διατυπωθεί, περιορίζει επίσης το δικαίωμα ασύλου, όπως να σε επαφή με αρχές τρίτου της χώρας για τα άτομα τα οποία κινδυνεύουν από διώξεις. Ε, σε ό,τι αφορά την περίοδο εθελοντικής επιστροφής, ε, εδώ υπάρχει απόλυτη απαγόρευση τέτοιας περιόδου ή προποθέσει και αυτό είναι πρόβλημα. Δεν, δεν μπορεί να ακουστεί δηλαδή η, η άποψη του ενδιαφερομένου δεν υπάρχει μια δυνατότητα ένδικων μέσων είναι πολύ περιορισμένο το χρονικό διάστημα ε, για να προσφύγει κάποιος έτσι λοιπόν εδώ κινδυνεύει και η αρχή της μη ε, απόκρουσης ε, είναι δύσκολο να αξιολογήσουμε τώρα ε, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία στα σύνορα ε, ποιο είναι ο αντίκτυπο, διότι αυτό εξαρτάται και από τι συζητήσει που λαμβάνουν στα πλαίσια του, του κανονισμού για το άσυλο. Τώρα μα θέσετε και ένα ερώτημα ε, σχετικά με την συνέπεια σε σχέση με άλλα νομοθετήματα τη ε, Ένωση στον συγκεκριμένο τομέα. Πάλι μιλάμε για εστιασμένη μελέτη αντικτύπου, εξετάσαμε δηλαδή μόνο ε, αυτή την πρόταση σε σχέση με κάποια νομοθετήματα και αυτό οδήγησε σε δύο σχόλια. Πρώτα απ' όλα διαπιστώσαμε ότι αυτό που είναι εντυπωσιακό στην πρόταση αυτή, ότι είναι μια σειρά από διατάξεις, δημιουργούν όχι μόνο ένα ε, χαμηλό επίπεδο, ένα ελάχιστο επίπεδο προστασία, αλλά και ένα μέγιστο επίπεδο προστασία των δικαιωμάτων. Και αυτό είναι κάτι που ο νομοθέτη θα πρέπει να το προσέξει. Ε, θα πρέπει να το σκεφτεί δηλαδή. Και το δεύτερο σχόλιο έχει να κάνει με το γεγονό ότι ο περιορισμό ε, στι δικλείδε ασφαλεία, στι διαδικαστικέ, ε, για να προσφύγει κάποιο κατά μια απόφαση επιστροφή για κάποιον που έχει υποβάλει αίτημα διεθνού προστασία, όταν έχει απορριφθεί αυτό το αίτημα, ε, μπορεί το άτομο αυτό να έχει δικαίωμα προσφυγή και αυτό εδώ δεν του παρέχεται. Θα πρέπει λοιπόν να το προσέξουμε. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον συνάδελφο, νομίζω, τον δόκτωρα Φερνάντε, Την κυρία Φερνάντε, την δόκτωρα Φερνάντε. Ευχαριστώ. εγώ θα σας μιλήσω για τις οικονομικές επιπτώσεις αυτής της αναδιατύπωσης που προτείνεται. Ξεκινώντας με τη μεθοδολογία. Η αξιολόγηση έγινε στη βάση ορισμένων πηγών, ε, ερευνητικών, ε, από το δίκτυο μετανάστευσης, ε, αλλά και από έρευνες που, έχουν, που έχει διεξάγει ο IPRS στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης, αλλά και διάφορες αξιολογήσεις που έχουν γίνει από την Κομισιόν. Επίσης, ε, εξετάσαμε έρευνες που γίνονται σε τέσσερα κράτη-μέλη δεδομένου της εμπειρίας που έχουν συλλέξει κατά την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Γερμανία, Γαλλία, Τσεχία και Ιταλία είναι συγκεκριμένα τα κράτη-μέλη. Μάλιστα για αυτά τα κράτη-μέλη ζητήσαμε και κάποιες επιπλέον πληροφορίες στη βάση δεδομένων ασύλου και κάποιες πληροφορίες ε, μέσω ενό συγκεκριμένου κειμένου που του αποστήλαμε. Στην μας, αξιολόγησή μας ε, διακρίναμε δύο είδη κόστους και δαπανών. Ένα δηλαδή που αφορά το κόστος της αλλαγής των ε, των συστημάτων και δεύτερο ήταν οι οικονομικές επιπτώσεις που θα επιφέρουν αυτές οι αλλαγές όσον αφορά την κράτηση, την επικέντρωση σε αναγκαστικές και όχι πλέον οικειοθελείς επιστροφές κτλ. Όσον αφορά το άμεσο κόστος, διαπιστώσαμε ότι ε, κατοχυρώνονται σοβαρές ε, νέες δαπάνες και για τα κρατη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ε, συγκεκριμένα τέσσερα άρθρα, τα οποία και θα απαιτήσουν τις περισσότερες δυνατές αλλαγές τα 9, 14, 18 και 22. Τα κράτη-μέλη ε, θα χρειαστούν περισσότερες δαπάνες για την αύξηση του προσωπικού τους, για το συντονισμό των αρχών τους, των φορέων που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, την ε, υλοποίηση και πραγματοποίηση νέων μηχανογραφικών συστημάτων, αλλά και την ε, σύσταση νέων μονάδων στις αστυνομικές αρχές. Και τέλος, ε, υπάρχει και μια αύξηση του κόστους λόγω της αύξησης του αριθμού των ε, χώρων κράτησης αλλά και για τον ε, διαχείριση υποθέσεων ε, ανηλίκων κτλ. Επίσης, στην Ιταλία για παράδειγμα μάθαμε ότι 30 εκατομμύρια ευρώ έχουν προβλεφθεί για την οικοδόμηση νέων κέντρων κράτησης. Στο Βέλγιο ε, γίνεται ανακαίνιση κάποιων ε, χώρων υποδοχής και οικοδομούνται, κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή δύο επιπλέον. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο θα είναι το κόστος, αλλά πάντως είναι σίγουρα ένα κόστος το οποίο θα προκύψει από τη νέα οδηγία. Σε, Ευρωπαϊ... σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν τρία είδη κόστους. Ένα, ένα για την παρακολούθηση και τον συντονισμό, ένα κόστος για την ε, διεύρυνση του ρόλου της ΕΑΣΟ, άρθρο 18 και την ερμηνεία που δίνουμε εμείς στο άρθρο 22 και τέλος βλέπουμε και κάποιες επιπλέον ε, δαπάνες που σχετίζονται με την ε, αύξηση των οικειοθελών επιστροφών. Εδώ θα δείτε τα πορίσματα συνολικά, συμπερασματικά, στα οποία έχουμε καταλήξει και εδώ βλέπετε στις γραμμές πού ακριβώς θα υπάρξουν οι νέες δαπάνες, ανά άρθρο και τι είδους θα είναι αυτές οι οδηγίες. Από τα αριστερά προς τα δεξιά λοιπόν είναι οι περισσότερες κρατήσεις, λιγότερες ε, οικειοθελείς επιστροφές, περισσότερες ε, αναγκαστικές επιστροφές και διαχείριση αιτήσεων και ενστάσεων. Οι αναγκαστικές επιστροφέ ξέρουμε ότι κοστίζουν περισσότερο από τι οικειοθελεί επιστροφέ στα κράτη-μέλη. Άρα περισσότερες αναγκαστικές επιστροφές, περισσότερο κόστος. Γιατί χρειάζεσαι και περισσότερο προσωπικό για να τις επεξεργαστείς και να τις διεκπαιρέωσεις αυτές τις επιστροφές. Τα άρθρα 6, 7 και 22 λοιπόν οδηγούν ξεκάθαρα σε αύξηση των περιπτώσεων αναγκαστικής επιστροφής και ε, αυτό λοιπόν είναι το κόστος που προκύπτει από αυτή την μετάβαση, από, αυτή τη μεταστροφή από τις, αναγκαστικές, από τις οικειοθελείς στις αναγκαστικές επιστροφές και από την αύξηση των ενστάσεων που θα υποβληθούν. Επίσης, ε, αυξάνεται ε, ο αριθμός των παρανόμως διαμενόντων λόγω των νέων κανόνων και υπάρχουν και επιπτώσεις στην σκιώδη οικονομία. Ε, ωστόσο δεν καταφέραμε να ποσοτικοποιήσουμε και να μετρήσουμε επακριβώς τις επιπτώσεις αυτές ε, ως προς την οικονομική τους διάσταση. Όσον αφορά το κόστος της κράτησης, για να σας δώσω μια κλίμακα μεγέθους, εδώ βλέπετε ότι το επίπεδο το, της, του κόστους ε, ε στο χ βλέπετε τις, τους ισχύοντες κανόνες, το κόστος που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ενώ στον άξονα ψ βλέπετε την προβλεπόμενη αύξηση στις τέσσερις αυτές χώρες. Στα δεξιά βλέπουμε το Βέλγιο, 60 εκατομμύρια που είναι ακριβώς οι δαπάνες που αυτή τη στιγμή καταβάλλονται για ε, κράτηση, τα οποία και θα αυξηθούν στα 140 εκατομμύρια. Η Τσεχία είναι στο άλλο άκρο, αλλά και εκεί η ε, αύξηση του κόστους είναι πάρα πολύ μεγάλη, γύρω στα 2 εκατομμύρια. Αυτά από μένα αν έχετε ερωτήσεις, είμαι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, νομίζω ότι μπορούμε να ξαναδώσουμε τώρα το λόγο στην ε, εισηγήτρια για να υποβάλει τα σχόλιά της. Δεν ξέρω αν υπάρχουν συνάδελφοι που θα ήθελαν να θέσουν ερωτήσεις. Εγώ όμως έχω διαβάσει, μισοδιαβάσει αν θέλετε αυτές τις ε, εκθέσεις ε, πραγματικά είναι επώδυνο το να βλέπει κανείς πόσο είναι το κόστος. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που καταλήξατε και ε, συγκεντρώσατε όλα αυτά τα στοιχεία. Κάτι που μας δίνει ακόμη περισσότερους λόγους να δώσουμε έμφαση στην ε, οικειοθελή επιστροφή. Εκτός δηλαδή από τη διάσταση της αξιοπρέπειας των ανθρώπων, είναι και, έχει νόημα και από οικονομικής άποψης να δοθεί έμφαση και προτεραιότητα στις οικειοθελείς επιστροφές. Πρόεδρος. Μπάρμπαρα. Ήθελα απλώς να ευχαριστήσω για αυτήν την εξαιρετική μελέτη εντυκτύπου. Ένα σημείο με ενδιαφέρει όλος ιδιαίτερος και το έχω αναφέρει και στην προηγούμενη παρέμβασή μου. Τα δύο επίπεδα της εκδίκασης ή της λήψης απόφασης που αναφέρατε και στην ε, παρουσίασή σας, τα. Ε, διεπίπεδη δηλαδή δικαιοδοσία. Να μπορέσει κανεί να ασκήσει έφεση για μια απόφαση επαναπατρισμού. Αυτό που με ενδιαφέρει πολύ και θα ήθελα να μου πείτε είναι εάν γίνεται να έχουμε μια συνολική εικόνα του τι γίνεται στα κράτη-μέλη σε σχέση με την κατάργηση των δύο αυτών επιπέδων. Στην Ιταλία δεν υπάρχει αυτό το επίπεδο το διπλό, αλλά ένα μόνο. Νομίζω ότι και στη Γαλλία πήγανε στο ένα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποια είναι η κατάσταση σε άλλες χώρες, διότι φοβούμε ότι η ιδέα να έχουμε μια αποτελεσματική οδηγία για τους επαναπατρισμούς, για αποτελεσματικούς επαναπατρισμούς, τελικά η αποτελεσματικότητα θα καταλήξει ένα συνώνυμο της ταχύτητας. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ταυτόσιμη η δύο Ευχαριστούμε. Άλλες ερωτήσεις προς την ομάδα που εκπώνησε τη μελέτη. Υπάρχει κάποιος ε, από την ίδια τη μελέτη, κάποιος ε, ερευνητής που θα ήθελε να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή. Θέλω να είμαι σαφής. Υπό την νομοθεσία για τα θεμελιώδη δικαιώματα αρκεί ένα επίπεδο δικαιοδοσίας. Αυτό και μόνο ε, συνάδει με την σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν όμως κράτη-μέλη πράγματι όπου υπάρχουν πολλές δικαιοδοσίες. Κάναμε συνεντεύξεις με κάποιους ε, εργαζόμενους σε εθνικές αρχές ε, που ζήτησαν την ανωνυμία τους, όπου εξέφρασαν ανησυχίες ότι δεν θα το να μην υπάρχει δυνατότητα περισσότερων επιπέδων δικαιοδοσία θα μπορούσε να δημιουργήσει συνταγματικά προβλήματα. Δεν έχω εξαντλητική εικόνα του αριθμού των επιπέδων δικαιοδοσία ε, στα κράτη-μέλη που θα μπορούσαν να πληγούν από αυτήν την νέα οδηγία. Δεν έχω αυτό το στοιχείο, αλλά σας διαβεβαιώ ότι πρώτον, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν θέλουμε θεμελιώδη δικαιώματα, δεν απαιτεί παραπάνω από ένα επίπεδα όμω όμως υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία έχουν ε, εκφράσει ανησυχία ότι θα έχουν συνταγματικά προβλήματα αν από την οδηγία απαγορεύεται να υπάρχουν πάνω από ένα επίπεδο δικαιοδοσίας. Ωραία. Λέω πρόεδρο. σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ε, μελέτη αντικτύπου και για την ποιότητα της δουλειάς σας. Θερμές ευχαριστίες σε ολόκληρη την ομάδα, λοιπόν, από εμάς. Έχουμε μια εξαιρετική εισηγήτρια, πολύ καλούς σκιώδεις, έμπειρους σκιώδεις και νομίζω ότι και με τη βοήθεια αυτής της μελέτης αντικτύπου θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα πολύ καλό θετικό αποτέλεσμα στο φάκελο αυτό. Είπα, έχουμε τους, την καλύτερη εισηγήτρια και την, ε, τους καλύτερους σκιώδεις σε αυτό το θέμα. Σας ε, παρατρύνω λοιπόν και εγώ να αξιοποιήσετε αυτές τις εξαιρετικές πληροφορίες που συνέλεξαν οι συνάδελφοι για εμάς. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ Judith και όπως είπαμε θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να συζητήσουμε το θέμα αυτό και με την Κομισιόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Κομισιόν και για τη δική σας συμβολή. Λοιπόν, αυτά και μπορούμε να περάσουμε στον Κοινοτικό Κώδικα Θεωρήσεων. Ο Χουάν Φερνάντο είναι εδώ. Μιλάμε για τον τελευταίο τριμερή διάλογο για τον κώδικα θεωρήσεων που έγινε σήμερα το πρωί Περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία να μας πει τι έγινε, τι διεμήφθη στον τριμερή διάλογο αυτόν σε σχέση με τον κώδικα θεωρήσεων. Χωάν Φερνάντο, έχει το λόγο. Να σας πω τι γίνεται. Μετά από τετραετής διαπραγματεύσεις με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, καταφέραμε σήμερα μόλις να καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία για τη διατύπωση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κώδικα Θεωρήσεων. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τους σκιώδεις συζητητές για όλη τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και που μας επέτρεψε να καταλήξουμε σε αυτή την ικανοποιητική λύση, έκβαση. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν στις τεχνικές συνεδριάσεις, δηλαδή τα μέλη της Γραμματείας και όλους τους βοηθούς. Ο αρχικός τριμερή διάλογος έγινε στις 14 Δεκεμβρίου υπό Αυστριακή Προεδρία. Στη συνέχεια κάναμε πάρα πολλές σοβαρές συναντήσεις σκιωδών τον Ιανουάριο, στι 9, στι 22 Ιανουαρίου που ακολουθήθηκαν από συναντήσεις τεχνικού χαρακτήρα και καταφέραμε να ε, συνοψίσουμε ε, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζαμε στις διαπραγματεύσεις. Επίσης, καταβάλαμε τεράστιες προσπάθειες για να καταλήξουμε σε ένα είδος γενικής συμφωνίας και συμφωνίας με ε, διάθεση συμβιβασμού που επέδειξαν και οι δύο συνομοθέτες. Κάτι που ήταν απαραίτητο για να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Μιλάω για την υποχρεωτική εκπροσώπωση με υποχρεωτικό συμβιβασμό με ρήτρα που θα εξασφαλίζει την καλύτερη εκπροσώπηση τα τέλη θεωρήσεων και παροχής υπηρεσιών, άρθρα 16 και 17, με γενική συμφωνία που σέβεται τα βασικά σημεία τα οποία ζητούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επί των οποίων συμφωνήσαμε την ε, θέση μας, καταλήξαμε σε συμφωνημένη θέση, την ε, προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων, άρθρο 19, σε πνεύμα συμβιβασμού, βάλαμε έξι μήνες με ειδική ε, πρόβλεψη 9 μήνυ για τους ναυτικούς και για 15 μέρες για την εξέταση ξεχωριστών ατομικών περιπτώσεων αλλά και την ε, ε, δυνατότητα ε, να καλεί την πίστη ταξιδιωτών να λαμβάνουν θεωρήσεις. Χρειάστηκε να ξεπεράσουμε κάποιες ε, ανησυχίες. Επίσης, στο άρθρο 8 υπάρχει μια ε, ρήτρα εγγύησης και υπάρχει και η διασύνδεση με την Κομισιόν. Εδώ καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα δύσκολο συμβασμό έπειτα από πρόταση διατύπωσης της Κομισιόν. Τη δυνατότητα δηλαδή να θεσπίζονται θετικά κίνητρα σε εκείνα τα, σε εκείνα τα κράτη που δείχνουν προθυμία ε, συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πολιτική επανεισδοχής. Και μετά υπάρχουν και τα, ε, το ζήτημα της ιατρικής ασφαλιστικής κάλυψης, άρθρο 15. Εδώ δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι θεωρήσεις ε, βραχίας διάρκειας δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στην βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και ιατρικής περίληψης των κρατών μελών. Ωστόσο, παρόλα αυτά, στο πακέτο τελικά θα περιλαμβάνεται σχετική διάταξη ε, για την ασφαλιστική ιατρική κάλυψη με ρήτρα αναθεώρησης όμως η οποία προβλέπει ότι πολύ σύντομα τα κράτη-μέλη θα υποχρεωθούν να υποβάλουν συγκεκριμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν την ε, δυσβάστακτη επιβάρυνση των κοινωνικών του συστημάτων, συστημάτων ασφάλισης και στη βάση αυτών των στοιχείων η Κομισιόν θα προβεί σε ενδελεχή ανάλυση και να δει, να δούμε από κοινού δηλαδή, αν θα διατηρηθεί αυτή η αρχή, αυτή η διάταξη ή αν θα καταργηθεί αυτή η διάταξη περί ταξιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης. Τέλος, τέλος υπήρξε και το θέμα των, ε, της υποβολής αιτήσεων ε, θεώρησης στα σύνορα από την πλευρά του Κοινοβουλίου υπήρχε αυτή η πρόταση. Το Συμβούλιο αντέδρασε στεναρά όμως στην θέσπιση ενός τέτοιου ε, καθεστώτος ε, και έτσι αναγκαστήκαμε για λόγους συμβιβασμού να αποδεχθούμε αυτή τη θέση του Συμβουλίου. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι αυτά τα τέσσερα χρόνια συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις, στις πολύ δύσκολες. Νομίζω ότι καταλήξαμε σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ανταποκριθήκαμε στο ρόλο μας και στην, στο καθήκον μας ως συνομοθετών να θεσπίσουμε νομοθεσία για τις θεωρήσεις, η οποία θα είναι επικαιροποιημένη ε, και θα συνάδει πλέον με τη συνθήκη της Λίσαβόνας και σε τελική ανάλυση Φυσικά η λύση που βρέθηκε δεν είναι 100% ικανοποιητική για όλες τις πλευρές. Συνολικά όμως νομίζω ότι μπορώ να πω ότι πρόκειται για ένα deal, μια συμφωνία συμβιβαστική και στο πλαίσιο αυτό με ταπεινότητα θα ήθελα να σας καλέσω να υποστηρίξετε αυτές, αυτούς τους συμβιβασμούς στους οποίους καταλήξαμε ώστε επιτέλους να τεθούν σε ισχύ τα όσα συμφωνήσαμε σε σχέση με τον κώδικα θεωρήσεων. Ευχαριστώ κύριε Μπέκερ, θέλετε να, να πείτε κάτι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, ο οποίος με πολύ μεγάλη θέρμη, αλλά και με συνέπεια, με την ομάδα του αλλά και με τη γραμματεία, κατάφερε να ε, επιτελέσει ένα πολύ σημαντικό έργο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδεις που με τα δικά τους επιτελεία ε, ε, συμμετείχαν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Χθες μόνο διήρκεσαν 7 ώρες Θέλω λοιπόν να συγχαρώ όλους όσοι συμμετείχαν για την ολοκλήρωση αυτού του τριμερούς διαλόγου. Για εμένα και για το ΕΛΚ είναι σημαντικό το γεγονός ότι εξασφαλίσαμε την ε, απλοποίηση των διατάξεων για ε, ερευνητές, αθλητές, ε, δημιουργούς, καλλιτέχνες ε, για τις επιχειρήσεις και αυτό είναι σημαντικό και είναι σημαντικό το ότι αυτό συνδυάζεται, πλέον με την ενισχυμένη συνεργασία με τις ε, τρίτες χώρες. Ότι δεν θα υπάρχουν θεωρήσεις στα εξωτερικά σύνορα, ότι διατηρήθηκε υποχρέωση για την ιατρική περίθαλψη, ε, ιατρική κάλυψη και όπω είπε και ο εισηγητή, βεβαίω θα υπάρξει μια αξιολόγηση όλων αυτών, αλλά αυτή τη στιγμή παραμένει η υποχρέωση ασφαλιστική κάλυψη ε, και νομίζω υγειονομική κάλυψης και νομίζω ότι ε, όλα αυτά αποτελούν ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα μια πολύ μακρά και δύσκολη διαπραγματεύση. Νομίζω ότι είμαστε ενώπιον μια πάρα πολύ σημαντική και θετική στιγμή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την Επιτροπή Ατομικών Ελευθεριών. Ευχαριστώ πολύ. Χουάν Φερνάντο για τη δουλειά σου, την πολύ σκληρή και περιμένουμε να δούμε το θέμα αυτό και στην Ολομέλεια τον Μάρτιο και από εκεί και πέρα αυτά. Συγχαρητήρια και από εμένα. Um, λοιπόν, να προχωρήσουμε στο σημείο 6 η διαδικασία σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο απόφαση του Συμβουλίου που καλεί τα κρατημέλη να προσχωρήσουν στην Σύμβαση για την Ολοκληρωμένη Ασφάλεια και τι υπηρεσίε που τα παρέχονται για ποδοσφαιρικού αγώνε και άλλε αθλητικέ εκδηλώσει του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Θα πρέπει να κυρωθεί η σύμβαση αυτή, ιδίω στα τμήματα αυτή που είναι αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υπογραφή και κύρωση τη σύμβαση από τι 3 Ιουλίου 2016 και σκοπό έχει να δημιουργήσει ένα ασφαλέ, προστατευμένο και ευχάριστο περιβάλλον για του ποδοσφαιρικού αγώνε και τι άλλε αθλητικέ εκδηλώσει. Θα δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στην κυρία Κάουφμαν. Θέλεις το λόγο, Σιλβί, για να παρουσιάσεις την έκθεσή σου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ποιο είναι το θέμα της έκθεσης. Συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης για, για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις. Η Συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης τέθηκε προς υπογραφή τον Ιούλιο του 2016. Και αυτή η συμφωνία είναι η μοναδική ε, σχετική διεθνή συμφωνία δεσμευτικού νομικού χαρακτήρα για την δημιουργία ενός μηχανισμού συνεργασίας μεταξύ όλων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που συμμετέχουν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο στην διοργάνωση ε, αθλητικών και πιο συγκεκριμένα ποδοσφαιρικών ε, διοργανώσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως δεν είναι συμβαλόμενο μέρος, ούτε μπορεί να είναι. Τα κράτη-μέλη της όμως μπορούν να είναι Κάποια όμως ε, ε, θέματα αυτής της συμφωνίας, ε, για κάποια μάλλον από αυτά τα θέματα που περιλαμβάνει η συμφωνία, χρειάζεται εξοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα άρθρα 2 έως 4 που αφορά τις τις, τα σημεία πληροφόρηση για το ποδόσφαιρο. Εδώ, σε επίπεδο ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει η απόφαση 348 του Συμβουλίου του 2002 για τους πεθασφαιρικού αγώνες που άπτεται των ίδιων θεμάτων. Εκείνοι λοιπόν που ε, συμμετέχουν ή παρακολουθούν ποδοσφαιρικούς αγώνες ή άλλες αθλητικές διοργανώσεις θα πρέπει να είναι ασφαλείς και να μπορούν να απολαμβάνουν ένα ευχάριστο περιβάλλον. Για αυτόν τον σκοπό λοιπόν χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις ε, για την παροχή απορρισιών, την προστασία της σωματικής ακαιρεότητας και την ασφάλεια. Με αυτόν τον τρόπο ε, προστατεύονται εκείνοι που θέλουν να παρακολουθήσουν αγώνες τόσο κατά το ταξίδι τους προς το σημείο διοργάνωσης ε, του αγώνα αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα στις εγκαταστάσεις της αθλητικές. Τις αθλητικές. Αυτό συνδέεται και με την ε, ε, ορθή συμπεριφορά που πρέπει να έχουν οι συμμετέχοντες και οι θεατές αυτών των οργανώσεων και να προβλέπονται συγκεκριμένε κυρώσεις σε περίπτωση βίας συμπεριφοράς. Πρέπει το περιβάλλον στα γήπεδα, στους ε, χώρους όπου διεξάγονται οι αγώνες να είναι ασφαλές ε, και να προστατεύει ε, παιδιά, ευάλωτους, γυναίκες, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να απολαμβάνει τέτοιου είδους αθλητικές διοργανώσεις. Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα παρακολουθεί την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και εδώ νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι δεν θα πρέπει να συμμετέχουν μόνο η UEFA, η FIFA και άλλοι ε, μεγάλοι ποδοσφαιρικοί, ε, ποδοσφαιρικές οργανώσεις αλλά ε, και οργανώσεις των οπαδών, των φιλάθλων. Εγώ υποστηρίζω τα διάφορα μέτρη, μέτρα που περιλαμβάνονται στο κείμενο για την εφαρμογή αυτή τη συμφωνία. Θέλω όμω να επισημάνω ένα συγκεκριμένο θέμα. Χαιρετίζω το γεγονό ότι η συμφωνία περιλαμβάνει την προσέγγιση ότι τα συμβαλόμενα μέρη σε περίπτωση ρατσιστικών ή σεξιστικών ή ομοφοβικών εκδηλώσεων στι ε, αθλητικέ διοργανώσει θα πρέπει να καταρτήσουν συγκεκριμένε κατευθυντήριε γραμμέ για την καταπολέμηση αυτών αλλά και για την απαγόρευσή του. Για μένα είναι απαραίτητο τα κράτη-μέλη να δώσουν ιδιαίτερη συμφωνία στην εφαρμογή αυτή της διάστασης. Η ανοχή, ε, το fair play, ο σεβασμός πρέπει να είναι στοιχεία που θα καθορίζουν και θα χαρακτηρίζουν και τις αθλητικέ διοργανώσεις αλλά και την κοινωνία μας συνολικά. Ελπίζω και σας παρατρύνω ως Κοινοβούλιο να υποστηρίξουμε αυτή τη συμφωνία, αυτή την εξουσιοδότηση προς τα κράτη-μέλη, ώστε να υπογράψουν αυτή τη συμφωνία και βεβαίω θέλω ε, από αυτό το βήμα να καλέσω βεβαίω και τα κράτη-μέλη το συντομότερο δυνατό να προχωρήσουν στην κύρωση αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστούμε, Σιλβί Βόν για τι εξηγήσει σου. Πολύ ενδιαφέρουσα η όλη διαδικασία. Και για το τι γίνεται με του ποδοσφαιρικού αγώνε. Εγώ θυμάμαι ότι ήσουν αντιπρόεδρο όταν καταφέραμε να εγκριθεί η πρώτη γραπτή δήλωση για τον αυξανόμενο ρατσισμό και την επανεμφάνισή του στου αθλητικού αγώνε στα ποδοσφαιρικά μάτ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήσουν εσεί η γήτρια και καταφέραμε να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Ήταν επιτυχία για μα. Σημαντικό λοιπόν. Πρώτη δήλωση για το θέμα αυτό. Δεν ήταν εύκολο να συλλέξουμε τις ε, απαραίτητες υπογραφές. Το θυμάμαι ακόμα. Συνάδελφοι, κάποιος από τους Κιώδης θα ήθελε το λόγο. Κύριε Σόγκορ. Με συγχωρείτε που πετάχτηκα. Είναι τρίτη απόγευμα. Παρακαλώ για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, δεν πειράζει. Σας δείχνουμε κατανόηση. Ε, βρετανικό ποδόσφαιρο. Παραμείνετε ευγενεί παρακαλώ. Δεν είμαι υποστηριχτή των αγγλικών ομάδων, αν και είμαι των σκοτσέζικων. Τέλο πάντων, α μην μπούμε τώρα σε αυτέ τι λεπτομέρειε. Ναι, Ευχαριστώ. Ε, συμφωνώ με το σκεπτικό να επικαιροποιηθούν οι κανόνες του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις περιπτώσεις βίας σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και αθλητικές εκδηλώσεις. Το να έχουμε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας στον τομέα αυτό δεν αρκεί όπως στο παρελθόν. Πρέπει να έχουν την ευχαριστότερη δυνατή εμπειρία όσοι παίρνουν μέρος στις αθλητικές εκδηλώσεις. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει τάξη, ασφάλεια και προστασία ώστε όλοι να μπορούν να ευχαριστηθούν την αθλητική εκδήλωση των αγώνα. Ε, υπάρχουν κάποιες ε, προσφυγές για εκφράσεις ρατσιστικές, εκφράσεις μίσου, αυτές αμαυρώνουν πολλούς αθλητικούς αγώνες. Υπάρχει και περίπτωση κακοποίησης παικτών από τη χώρα με την Ρουμανία, ας πούμε, έχουμε δει τέτοιες περιπτώσεις και αναφέρονται και τις εκθέσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για αυτό και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και του κανόνε τη Σύμβαση για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων. Τέτοια συμπεριφορά δεν μπορεί να γίνεται δεκτή σε ποδοσφαιρικά ε, στάδια αθλητικά και οποιαδήποτε βίαιη συμπεριφορά κατά της ουγγρικής μειονότητας ε, δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτή ή εκφράσεις μίσους. Φυσικά ακόμη και αν αυτά δεν καταλήξουν σε βία επεισόδια στο στάδιο, στο, γήπεδο μπορεί να προεκταθούν εκτός του αγώνα αμέσω μετά. Θα πρέπει λοιπόν η ανεκτικότητα, ο σεβασμός, η δίκαιη διεξαγωγή του παιχνιδιού να είναι αρχές που θα διέπουν όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις όσο το δυνατόν περισσότερο. Γι' αυτό είμαστε υπέρ της εναρμόνισης των προτύπων και της ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα αυτό. Καλωσορίζουμε τη νέα σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη-μέλη να υπογράψουν και να κυρώσουν όσο το δυνατόν συντομότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σόγκορ. Ενδιαφέρον. Κύριε Γιούρεκ, και εσείς είστε σκιώδης, θέλατε το λόγο. Νομίζω αυτά είναι όλα για τους περισσότερους από τους συναδέλφους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να μας πει κάτι. Κύριε Γιωτάκος, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή καλωσορίζει το σχέδιο σύμβασης του Συμβουλίου που έχει υποβάλει ο εισηγητής. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε τη δυνατότητα να ευχαριστήσουμε και την Επιτροπή ΚΑΛΤ για τη θετική της προσέγγιση από τις 2 Ιανουαρίου για το θέμα αυτό και τώρα εφόσον έχει υποβληθεί το σχέδιο κανονισμού ε, περιμένουμε τη συμφωνία γνώμη του Κοινοβουλίου ώστε το Συμβούλιο με τη σειρά του να μπορέσει να εγκρίνει και τυπικά την απόφαση. Η διαδικασία κύρωσης θα ξεκινήσει αμέσως, τέλος πρώτων θα συνεχιστεί ή θα ξεκινήσει με τη σωστή νομική βάση, για να το πω καλύτερα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι όπως υπόθηκε και κατά τη διάρκεια της συζήτησής σας, για το σχέδιο σύστασης. Καλό είναι να αποσαφινιστεί η νομική κατάσταση για τα κράτη-μέλη που είναι και μέλη και έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Από το Συμβούλιο, η Προεδρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο. Για το θέμα αυτό μπορούμε να πούμε ότι και εμείς καλωσορίζουμε την όλη συζήτηση. Είναι πολύ θετικό το σχέδιο έκθεση. και το ίδιο και οι εξηγήσει τη εισηγητρία. Το ξεκινήσαμε στην ε, ομάδα εργασία για την ενίσχυση του δικαίου τον Ιούνιο. Είχαμε και τη σχετική γνωμοδότηση τη νομική μα υπηρεσία. Έχουμε υποβάλει το θέμα στο Κορέπερ και το Συμβούλιο από τον Οκτώβριο. Οπότε ζητούμε την σύμφωνη γνώμη σας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην έγκριση της απόφασης η οποία θα γίνει μόλις λάβουμε τη σύμφωνη γνώμη. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ που προβλέψατε αυτό το θέμα προς συζήτηση και απλώς να πω ότι το Συμβούλιο θα προχωρήσει αμελητή ε, μόλις ε, ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Ευχαριστούμε και τώρα εισηγήτρια και πάλι. Λιβόν. Ευχαριστώ Κλοντ και ε, σε ευχαριστώ και για το γεγονό ότι υπενθύμησε στην, τον επίγοντα χαρακτήρα της πολιτικής κατάστασης. Όποτε έχουμε παγκόσμια πρωταθλήματα ποδοσφαίρου ή ευρωπαϊκά ε, πρωταθλήματα ε, με αυτές τις ε, ε, εκστρατείες κατά του ρατσισμού ε, θυμάμαι ότι το Κοινοβούλιο ήταν από τους πρώτους που έθεσαν αυτό το θέμα στην ε, δημοσιότητα, στην επικαιρότητα. Όποτε λοιπόν γίνονται τέτοιες εκστρατείες αντιρατσιστικές, ε, νομίζω ότι πραγματικά πρόκειται και για μια διαδικασία στην οποία έχουμε συμβάλει και εμείς. Γιατί ο ρατσισμός ειδικά στον αθλητισμό είναι τεράστιο πρόβλημα γι' αυτό και ε, χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι κατέληξε το Συμβούλιο της Ευρώπης σε αυτή την εξαιρετική συμφωνία πρέπει και εμείς λοιπόν να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μας στο συντομότερο δυνατό για να μπορέσει να ξεκινήσει η σχετική δουλειά να πω κάτι για τις προθεσμίες συγκεκριμένα θέλουμε στις 19 Φεβρουαρίου να γίνει η ψηφοφορία εδώ στην Επιτροπή και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει στην πρώτη Ολομέλεια του Μαρτίου. Ευχαριστούμε, Σιλβί Θα αποβληθούν τροπολογίες μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για αυτή την πολύ θετική παρουσίαση. Σημείο 7 τώρα. Το θέμα για την πρόταση της διευκόλυνσης για τη χρήση οικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, ε, έρευνα και εντοπισμό ή δίωξη κατά κάποιων ποινικών αδικημάτων. Είναι στο τελικό στάδιο η όλη η διαδικασία διαδικασια υποματρεψης με δύο γύρου τριμερών διαλόγων, τεχνικέ συνεδριάσεις... και αυτό μετά την ανακοίνωση τη εντολή, την έγκριση μάλλον τη εντολή από την Ολομέλεια του Δεκέμβρη. Ο εισηγητή είναι ο κύριο Ράντεφ. Βλέπω ότι έχει καταφτάσει, οπότε κύριε Ράντεφ, παρουσιάστε μας το πώς έχουν προχωρήσει οι διαθεσμικέ διαπραγματεύσει για το θέμα σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Θα είμαι πολύ σύντομος. Η όλη διαδικασία για την έγκριση του, του θέματος αυτού ήταν ε, πολύ εντατική. Είχαμε δύο γύρους τριμερών διαλόγων και πολλές τεχνικές συνεδριάσεις από το Δεκέμβριο. Έχουμε, έχουν δουλευτεί ήδη πολλά τμήματα του κειμένου, αλλά υπάρχουν και κάποια εκκρεμή. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει αρκετέ προτάσει για να καταλήξουμε σε συμβαστικέ λύσει για το θέμα αυτό. Οι συμβαστικέ όμω απορρίφθηκαν από τα κρατη Έχουμε έναν ακόμα γύρο τριμερούς διαλόγου και εάν θέλουμε το όλο θέμα να εγκριθεί ως το τέλος της θητείας, δεν έχουμε πλέον πολύ χρόνο. Εάν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ένας ασφαλέστερος χώρος ανταλλαγής πληροφοριών, θα είμαι σαφής. Ε, οι συμβαστικές λύσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου θα πρέπει να περάσουν. Ιδάλλως δεν θα υπάρξει συμφωνία και θα έχουν την ευθύνη τα κράτη-μέλη μόνα του. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι η ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να συνεχιστεί ως έχει. Δεν είναι κατάλληλο το επίπεδο ανταλλαγή πληροφοριών τώρα. Χρειάζεται αναβάθμιση, χρειάζεται βελτίωση με τόσε τρομοκρατικέ απόπειρε και τι διασυνδέσει ε, του, οικονομικού, του οργανωμένου εγκλήματο με τα δίκτυα που το χρηματοδοτούν. Ευχαριστούμε, κύριε Ράντεφ. Ευχαριστούμε πολύ κιόλα. Κάποιες φορές ωραία θα ήταν να μιλάγατε λίγο παραπάνω. Έχουμε προγραμματίσει ψηφοφορία στις 4.30. Κάποιες φορές εύχομαι να είχαμε πιο πολλές ψηφοφορίες για να τελειώνουμε, αλλά θα ζητήσω συγγνώμη, διότι θα ήθελα να έχουμε οργανώσει διαφορετικά το πρόγραμμα για να μην χάνετε κι εσείς το χρόνο σας. και ούτω ή άλλω κάτι θα πρέπει να αναβληθεί για την επόμενη Δευτέρα. Οπότε συγγνώμη που σε έφερα εδώ. Μία ψηφοφορία μόνο έχουμε. Ζητώ συγγνώμη. Δεν αλλάζει τίποτα προ το καλύτερο επειδή είναι δική μου η έκθεση. Πάντως ευχαριστώ για την προσέλευσή σας και θα ξεκινήσουμε Ε, θα ξεκινήσουμε μόλι έρθουν και άλλοι συνάδελφοι που θα του δείξουμε λίγο σεβασμό και θα του περιμένουμε γιατί θα έρθουν μόνο για αυτή τη μία ψηφοφορία. Οπότε θα κάνουμε ένα διάλειμμα για πέντε λεπτά αν δεν σα πειράζει, εντάξει, παρά που κάποια από εσά ήδη ήρθατε. Τι έγινε, αποκοιμηθήκατε. Δεν ξέρω αν η φωνή μου σα να νουρίζει. Um, okay, don't laugh too loud because that's not very nice. But um, Yes, see, people are coming in for this vote, so can we pause for five minutes? Μπορούμε να κάνουμε πέντε λεπτά διάλειμμα και μετά θα ψηφίσουμε. Okay. Okay, we pause for five minutes. Πέντε λεπτά διάλειμμα και θα ψηφίσουμε. I'm very sorry. It's a little bit inconvenient for everyone, but we'll do that.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 Um, Συνάδελφοι, απλώς να σας πω ότι εάν έχετε έρθει για τις προφορίες και θέλετε να φύγετε, μη φύγετε, χρειαζόμαστε ενισχυμένη πλειοψηφία. Αν είστε εδώ λοιπόν για να ψηφίσετε, παρακαλώ περιμένετε, μείνετε. Χρειάζεται ενισχυμένη πλειοψηφία για αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ.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

για Uh, um, Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ πάρτε θέσεις για να ψηφίσουμε. Λοιπόν, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη πρώτα απ' όλα που σας έφερα εδώ όλους για μια ψηφοφορία. Σκοπεύαμε να έχουμε και άλλοι για να έχει νόημα να είστε εδώ. Όμως ε, αναβλήθηκε μια ψηφοφορία για τη Δευτέρα και αυτό είναι κάτι το οποίο, για το οποίο δεν ευθυνόμαστε. Ε, πάντως, συγγνώμη που ήρθατε μέχρι εδώ για μία μόνο ψηφοφορία. Ψηφίζουμε λοιπόν ε, και πρέπει να ψηφίσουμε αυτό το θέμα σήμερα, διότι πρέπει να γίνει ανακοίνωση στην Ολομέλεια 30 Ιανουαρίου και αν δεν ψηφίσουμε σήμερα, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν μπορεί να συμβεί και εκτιμούμε ιδιαίτερα που ήρθατε για την ψηφοφορία αυτή. Ευχαριστώ για το χρόνο σας και την υπομονή σας να προχωρήσουμε. Ε, ειδική πλειοψηφία χρειάζεται, μην το ξεχνάτε, για την τελική ψηφοφορία κυρίως. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Υπάρχει και ένα διαδικαστικό ζήτημα από ό,τι, ξέρω, το οποίο έχει θέση να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία όμως πρώτα. Yeah, but then we start the vote and then she presents the oral amendment. Yeah, then we start the vote. Okay, so I'm starting the vote. Αρχίζουμε λοιπόν την ψηφοφορία. Ε, ζητώ την επικιά σας, έτσι. Ξεκινούμε την ψηφοφορία. Υπάρχει πρόταση για προφορική τροπολογία. Μάλεν, έχεις πρόταση προφορικής τροπολογίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαιρόμαστε που έχουμε έρθει εδώ να ψηφίσουμε. Μην ανησυχείτε. Προφορική τροπολογία λοιπόν για την κατάσταση στην Ιεμένη είναι η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο. Έχουν πάρει θέση στην Ολομέλεια για την αύξηση ε, της πίεσης προς την Σαουδική Αραβία και δεν υπάρχει κανένας, καμία νόμιμη οδός για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να βρεθούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική αυτή η τροπολογία. Ζητούμε δράση για τους Ιεμενίτες αλλά και για τους υπόλοιπους. Χρειάζονται ανθρωπιστικές θεωρήσεις για αυτούς. Δεν μπορεί να περιμένει αυτό. Γι' αυτό θέσαμε αυτή την προφορική τροπολογία. Όπως αντιλαμβάνεστε το περιεχόμενο αυτού που είπες ε, ε με βρίσκει σύμφωνο όμως σε ό,τι αφορά την προφορική τροπολογία υπάρχει ένα ζήτημα του κατά πόσο δηλαδή εμπίπτει στη συγκεκριμένη έκθεση. Επ' αυτής της βάσης λοιπόν ως εισηγητής ε, ε θεωρώ ότι δεν ταιριάζει σε αυτήν την, ε, ε, στην έκθεση παρότι συμφωνώ με το περιεχόμενο θα ήθελα να ξέρω αν έχει κάποιος αντίρρηση για αυτή την προφορική τροπολογία. Ναι, παρακαλώ τέσσερις αντιρρήσεις. Βλέπω παραπάνω από τέσσερις. Λοιπόν, ε, το περιεχόμενο λοιπόν έχει τη συμπάθειά μου, αλλά αφού υπάρχουν πάνω από τέσσερι εντηρήσει, δεν μπορούμε να ε, συμπεριλάβουμε αυτή την προφορική τροπολογία. Πάμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 12. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται και αυτή εκτιμώντας τώρα τροπολογία 1. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία απορρίπτεται τροπολογία 2 συγγνώμη τροπολογία 3 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται συμβασμός 1 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Τροπολογία 10. η ψηφοφορία. Ναι, είμαι αργός και νευρικός σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Πέρας ψηφοφορίας. Επειδή είμαι Βρετανός αυτό λέτε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Λοιπόν, τελική ψηφοφορία. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας με 53 ψήφους υπέρ 11 καμία κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Εγκρίνεται λοιπόν, υπερψηφίζεται. Χρειαζόμαστε και μια εντολή όμως, με ειδική πλειοψηφία. Παρακαλώ ψηφίστε και για την εντολή. Βλέπω, μάζεψε την κάρτα σου, Σιλβί, εγώ φταίω. Δεν έχουμε φύγει ακόμα, έτσι. Πέρας ψηφοφορίας, 50 υπέρ, 2 κατά. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας, συνάδελφοι. Μπορεί πλέον να πάει στην Ολομέλεια το θέμα. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη που ήρθατε και μόνο μία ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ευχαριστώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε εξέταση του σημείου 10, εάν ε, θέλετε. Κύριε Ντιόν, ζητώ συγγνώμη. Βεβαίω ε, υπάρχουν διάφορες, έτσι, διάφορα πηγατάκια. Ξεκινάμε την εξέταση του επόμενου σημείου, συνάδελφοι, Παρακαλώ, εάν θέλετε να συζητήσετε, βγείτε έξω. Συνεχίζουμε με την ημέρα διάταξη. Το επόμενο σημείο λοιπόν είναι η πρώτη πρόταση κανονισμού για την ε, ανταλλαγή προγραμμάτων συνδρομής ε, για την προστασία του ευρώ ε, από την παραχάραξη την περίοδο 2021-2027. Πρόκειται για το πρόγραμμα Περικλής Βόρ. αυτό αποτελεί μέρος του, του πολίτη δημοσιονομικού πλαισίου. Ο κύριος Διόν είναι ο εισηγητής. Όταν παρουσίασε το σχέδιο 6, θα θυμάστε στις 7 Ιανουαρίου ε, θα εξετάσουμε τώρα τις τροπολογίες. Έχουμε και μια τριανταριά τροπολογίες και 4 Φεβρουαρίου θα έχουμε την ψηφοφορία. Αναμένουμε λοιπόν να μάθουμε τι συμβαίνει με την έκθεση αυτή. Θα ακούσουμε τον εισηγητή. Ντένις, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Κλοντ. Είναι μικρός αριθμός των τροπολογιών, όπως είπες και εσύ. Είναι και ένα πρόγραμμα αρκετά ε, περιορισμένο. Το επικροτούν τους στόχους του προγράμματος όλοι οι σκιώδες ηγητής. Κανείς δεν θέλει ε, να υπονομευθεί η εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή οικονομία με πλαστά ευρώ. Ο στόχο λοιπόν του προγράμματο ε, δεν νομίζω να δημιουργεί πρόβλημα, δεν υπήρξε κάποια διαφωνία τουλάχιστον. Όσο το εξετάζω, τόσο αναρωτιέμαι κατά πόσο χρειάζεται ένα ειδικό πρόγραμμα βέβαια γι' αυτό, πέρα από το πρόγραμμα Justice. Υπάρχουν άλλοι τομεί στην ενιαία αγορά, όπου υπάρχει ένα πρόγραμμα για την ενιαία αγορά, Δεν το έθιξα όμως αυτό στην έκθεσή μου. Εμείς εργαστήκαμε επί τη βάση αυτού του προγράμματος ως ξεχωριστό πρόγραμμα και προσπαθήσαμε να ενσωματώσουμε όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία. Το βασικό στοιχείο που προκύπτει από τις τροπολογίες και πρέπει να, το συμπεριλάβουμε, πρέπει να συμπεριλάβουμε και τρίτες χώρες. Είτε χρησιμοποιούν το ευρώ, είτε έχουν πληροφορίες ε, για ε, δραστηριότητες ε, Επίσης η σχέση συνεργασίας με την Europol και την ECP ε, πρέπει να υπάρχουν οι δείκτες ε, απόδοσης οι οποίοι όμως πρέπει να είναι μετρήσιμοι χωρίς να δημιουργείται κάποιο διοικητικό άχθος. Σήμερα το πρωί λοιπόν είχαμε την πρώτη και μοναδική συνάντηση των σχεδόν εισηγητών την ερχόμενη εβδομάδα άλλωστε είναι η ψηφοφορία ήταν επικοδομητική η συνάντηση εντοπίσαμε τέσσερις ε, συμβαστικές τροπολογίες ε, για τους στόχους του προγράμματος ε, αλλά και την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε για τους δείκτες κλειδιά, δείκτες απόδοσης τελικά φτάσαμε σε κάποιους δείκτες που πραγματικά μπορούν να μας δείξουν ποια είναι η χρησιμότητα του προγράμματος γενικότερα για το ζήτημα του παραχάραξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τέλος ως εισηγητής έλαβα και μια επιστολή για το οριζόντιο ζήτημα των πράξεων κατεξιοδότηση αυτό αφορά όλα τα προγράμματα δεν είναι μια τροπολογία κάποιου όμως αν θέλουμε να ευθυγραμμιστούμε με τα άλλα προγράμματα υπάρχει πλέον μια συμβαστική πρόταση που προβλέπει ότι το πρόγραμμα εργασιών θα περάσει από πράξη κατεξιοδότηση όπως και τα υπόλοιπα προγράμματα. Εκεί λοιπόν βρισκόμαστε. Νομίζω ότι υπάρχει ευρεία συνένεση για αυτήν την προσέγγιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι πραγματικά ένα θέμα συναρπαστικό αυτό της παραχάραξης. Τόμα, εσύ ίσω και ο για το ΕΛΚ, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποστηρίξω ε, το θέμα αυτό. Είπε και ο συνάδελφος Ντένις Ντε Ιόγκ, ε, όταν προείδευσε εξαιρετικά την ε, συνάντηση σήμερα και πραγματικά ήταν τιμή μου που συμμετείχα σε αυτή τη συνάντηση των σκιών εισηγητών. Ήταν επικοδομητικό το κλίμα. Είχαμε μια πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων. Ορισμένε φορέ είναι αναγκαίο να μην υποβάλλονται πολλέ τροπολογίε ε, για ένα μικρό πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί και καλά. Ε, νομίζω ότι υπάρχουν τρία-τέσσερα σημεία συμβιβασμού ε, τα οποία υποστηρίζουν όλοι και πήγαν πολύ καλά τα πράγματα. Χαίρομαι που μεταξύ των ομάδων, των πολιτικών ομάδων, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια διαφωνία μεταξύ των σχεδόν εισηγητών. Θέλουμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε από κοινού ε, την εξέταση με μια μεγάλη συμβαστική λύση ε, που θα μας διευκολύνει στο μέλλον Πολύ μεγάλη υποστήριξη λοιπόν προς τον τένις ε, και συγχαρητήρια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συνεργάστηκα μαζί του γύρω από το έγγραφο αυτό. Άλλος κανείς θέλει το λόγο για το θέμα αυτό. Ωραία, ευχαριστώ Ντένις. Τέσσερις του μήνα ψηφίζουμε στην Επιτροπή. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Α, συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θέλει να μιλήσει για το θέμα αυτό. Δεν αφορά εμάς βέβαια αυτό. Εκοφίν Είναι το κομμάτι εκοφήν, έτσι, της Κομισιόν. Φαίνεται η διαφορά. Να είστε κάπως σύντομοι. Ναι, θα είμαι εξαιρετικά σύντομος. Εκπροσωπούμε την ε, Γενική Διεύθυνση ΕΚΦΙΝ που είναι υπεύθυνη για αυτό το πρόγραμμα, το Περίκλες. Έγινε μια πολύ καλή δουλειά από τον εισηγητή και του χιλιάδε εισηγητέ και εμεί ε, είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό. Υπάρχει ένα θέμα κλειδί για το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέλει να στήσει την προσοχή σα. Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα μικρό πρόγραμμα, όπω γνωρίζετε, και αποτελείται από ένα διαγωνισμό με δύο προθεσμίες εάν υπάρξει πράξη κατοξιοδότηση για να εγκριθεί το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών, αυτό θα δημιουργήσει πρώτα απ' όλα διοικητικό και δεύτερον ε, θα μας περιορίσει χρονικά διότι οι πράξεις όπως ξέρετε ε, περιλαμβάνουν μια δίμηνη περίοδο όσο το ολοκληρωθούν και είναι αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα βεβαίως θα πρέπει να λάβει χώρα διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τη Europol, τα κράτη-μέλη και αυτό παίρνει χρόνο, οπότε τελικά μπορεί να έχουμε ένα ετήσιο πρόγραμμα εργασιών το οποίο θα μπορέσει να εγκριθεί μόλις την Άνοιξη και αυτό είναι πρόβλημα πρώτα απ' όλα διότι ο οικονομικός κανονισμός αναφέρει ότι η αποφάση χρηματοδότησης ε, σύμφωνα με το άρθρο 1.110 του Κοριστατικού Κανονισμού πρέπει να εγκριθούν πριν τέλη Μαρτίου ε, οπότε και δεύτερον ε, θα δημιουργηθούν και προβλήματα για τους δικαιούχους διότι θα έχουμε μόνο μία προθεσμία για το διαγωνισμό το φθινόπωρο αυτό υπονομεύει κατά τη γνώμη μας την αποτελεσματικότητα του προγράμματος και δεύτερον, σύμφωνα με την νομική μας υπηρεσία, η έγκριση του πετήσιου προγράμματος εργασιών και η οικονομική απόφαση σχετική δίνει την, ε, μια αρμοδιότητα στην Κομισιόν να εφαρμόσει τον προπολογισμό με βάση το άρθρο 317 της Συνθήκης ε, και αυτό δεν μπορεί να ε, γίνει με μια πράξη κατοξιδότηση. Θα δούμε βεβαίω σε ποιο βαθμό θα μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με τους εμπλεκόμενους φορείς. Υπάρχει ήδη το άρθρο 4 για τη διαβούλευση και το, και 8 της πρόταση της Κομισιόν. Θα πρέπει να γίνει μια διευκρίνηση εκεί. Είμαστε διευθυμένοι να το κάνουμε. Όμως δεν βλέπουμε να υπάρχει προσταμένη αξία αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τι πράξει εξουδότηση, λαμβάνοντα υπόψη την ιδιαιτερότητα του προγράμματο, το μικρό προπολογισμό και του λίγου τελικά δικαιούχου. Ε, δεν νομίζω λοιπόν ότι εδώ χρειάζεται πράξη κατεξουδότηση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Thank you. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους από το ΕΚΟΦΗΝ. Αστειευόμουν προφανώς. Ε. Είναι πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθεί κανείς διαφορές ανάμεσα στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, το ΕΚΟΦΗΝ και τις διαφορετικές οπτικές που προσφέρει ο κάθε φορέας, το κάθε σώμα σε αυτά. Σας ευχαριστούμε λοιπόν όλους για τη συμμετοχή σας ε, στη συζήτηση αυτή και την όλη διαδικασία. Αυτά. Λοιπόν, θα κάνουμε πάλι ένα μικρό διαλυματάκι γιατί έχουμε προσκαλέσει την κυρία Γιούροβα, την Επίτροπο εδώ στις 5 είναι καθοδόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν τους συναδέλφους. Έχουμε ε, πολύ σημαντικά θέματα να συζητήσουμε μαζί της. Σας παρακαλώ μη φύγετε. Μας έχει πει ότι θα είναι εδώ στις 5. If you Thank you.

Uh, ε, συνάδελφοι, συγγνώμη, έχει αργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ξέρω γιατί. Οπότε δεν λέω ακριβώ συγγνώμη. Εδώ που τα λέμε, η Κομισιόν φταίει. Απλά σα ενημερώνω για το τι γίνεται. Okay, the commissioner is on her way and... Λοιπόν, είναι καθοδόν η Επίτροπος, αλλά πέραν αυτού δεν έχω ιδέα που ακριβώς είναι. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας ζητήσω συγγνώμη και να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας. Uh, Συγγνώμη, μίλησα μόλις με την Επίτροπο. Είχε πρόβλημα, έχει, έχουν ποτηλιαριστεί οι δρόμοι. Βρίσκεται όμως μπροστά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα είναι εδώ σε δύο λεπτά. Μόλις μπήκε στην είσοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έρχεται, τρέχει extra information. That's most helpful. Ευχαριστούμε για αυτές τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες. We should film this committee for like a kind of sitcom or reality TV show. Μήπως θα ήμασταν ε, καλή κομμυρική σειρά και να ήμασταν εμείς οι πρωταγωνιστές. Πλάκα θα είχε. Ευχαριστώ πάντως για τις πληροφορίες αυτές. Δύο λεπτά μας είπες, ε. calling me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 So that was the commissioner on the mobile, because I just want to continue with the kind of thing that Thomas has done to give your... Η Επίτροπος ήταν στο κινητό και θέλω να σας ενημερώνω real time, θα συνεχίσω αυτό που έκανε ο Thomas, Έρχεται. Σε δύο λεπτά. Υπήρξε ένα πρόβλημα. Keep you up to date, you know.

Um, Συνάδελφοι, έγινε μια μικρή παρεξήγηση μάλλον. Σας ευχαριστώ πάντως για την υπομονή σας. Ευχαριστώ και την Επίτροπο που είναι εδώ μαζί μας. Αντί λοιπόν να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες, νομίζω ότι καλύτερα θα ήταν να ξεκινήσουμε. Εντάξει, είναι και αργά ε, και περιμέναμε αρκετή ώρα με όλα αυτά πάση περιπτώσει, Επίτροπε, ξέρω ότι υπήρξε μια μικρή παρανόηση, μια παρεξήγηση σε σχέση με την ώρα που είχαμε πει. Τέλο πάντων, είχαμε μια, μια συνάντηση ε, εδώ για μια συζήτηση για την, ε, την ε, θέσπιση προγράμματος ανταλλαγών. Θέλουμε να μιλήσουμε για τις ηλεκτρονικές ενδείξεις, τα αποδεικτικά στοιχεία, να σας ε, υπενθυμίσω ότι η Επίτροπος ε, ήταν εδώ στην Επιτροπή μας και τον Οκτώβριο ε, και μας είχε πει τότε ότι για την ασπίδα ιδιωτικότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης είπα θα μας ενημέρωνε όποτε η τελική έκθεση θα δημοσιευόταν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν ε, κύριε Επίτροπε για τη διαθεσιμότητά σας, για την παρουσία σας, για τις επαφές που έχουμε έκτοτε μαζί σας όλο το διάστημα δηλαδή. Εγώ βήρα σας έλεγα εδώ και πέντε χρόνια. Βέρα μαθαίνω τώρα ότι σας λένε στην πραγματικότητα. Βέρα, λοιπόν, έχετε το λόγο και ε, ευθύ αμέσω θα γίνει και ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ Κλοντ, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. Να με συγχωρείτε που καθυστέρησα. Όταν ε, μου λέτε μια ώρα, φροντίζω να είμαι πάντοτε τυπική. Αλλά είχα σημειώσει στην ατζέντα μου 5,5. Λάθος προγραμματισμός. Με συγχωρείτε. Ε, απευθείας στο θέμα μας. Έρχομαι μετά την έγκριση της απόφασης ε, για την επαναπατρισμό. Γι' αυτό έρχομαι να σας ενημερώσω για την κατάσταση των πραγμάτων και για την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικότητας και για την προστασία των δεδομένων. Και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσω όλα τα θέματα που σας ενδιαφέρουν. Πρώτα απ' όλα για την ε, ασπίδα της ιδιωτικότητας και την σχετική αναθεώρηση. Ξέρω ότι και για εσά η αναθεώρηση των προσωπικών δεδομένων και τη προστασία του είναι μια από τι ψηλότερε πολιτικέ προτεραιότητε. Την περασμένη εβδομάδα μόλις με τον Ιάπωνα Πρωθυπουργό είχαμε συζητήσεις για την ε, σφαιρική και την παγκόσμια προστασία προσωπικών δεδομένων βλέποντας και το τι θα γίνει με την ε, τεχνητή ευθεία και άλλα τεχνολογικά βήματα. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε εδώ στο Κοινοβούλιο ότι σε διεθνές επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση όχι μόνο για να συμβάλλει στην όλη συζήτηση αλλά και για να ηγηθεί. Ε, έχουμε επιφέρει εμείς πολλές καινοτομίες, αλλά μπορούμε να προωθήσουμε και τα υψηλά μας πρότυπα. Για να πετύχει αυτό θα πρέπει να εμπνεύσουμε τους άλλους αντί να τους αποθαρρύνουμε, να τους βοηθήσουμε να κερδίσουν ξανά την εμπιστοσύνη τους, ε, αντί να φοβούνται και να είναι σε σύγχυση. Πραγματικά εδώ ε, είμαι πολύ περίεργη για τις ιδέες, του, Σε ό,τι αφορά τώρα τις πρόσφατες εξελίξεις, στις Βρυξέλλες ε, η δεύτερη αναθεώρησή μας δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2018 και εδώ είχαμε εταιρείε τη ιδιωτικότητα, ασπίδα ε, ιδιωτικότητα, διαβουλεύσει με τι κοινωνίε των πολιτών και από τι Αμερικανικέ αρχές τα σχόλια και τη συνεισφορά του. Επίση, οι Ευρωπαίοι φορεί προσφέρανε στην όλη διαδικασία στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με τις ΗΠΑ προφανώς έχουν ληφθεί υπόψη οι στο Κοινοβουλίο όπως εκφράστηκαν στο ψήφισμα του Ιουλίου 2018. Θα είναι κεντρική σημασία στο πώς θα διαπραγματευτούμε το θέμα με τις ΗΠΑ και τα αποτελέσματα που θα επιδιώξουν. Οι Αμερικανικές αρχές έχουν λάβει μια σειρά από βήματα για να ανταποκριθούν στις ερωτήσεις τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι ανησυχίε του ε, Κοινοβουλίου. Το Εμπορικό Μιλητήριο έχει, ε, μάλλον το Υπουργείο για τα εμπορικά θέματα, έχει φροντίσει να ακολουθήσει μια ενεργότερη ε, προσέγγιση για να ενισχύσει το πλαίσιο. τα μέλη του Συμβουλίου Εποπτείας για την ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων που δεν είχαν διοριστεί, τώρα έχουν διοριστεί και έχει ήδη δημοσιευτεί στις 28 γλώσσες σε σχετική ανακοίνωση στην επίσημη εφημερίδα. Έχουμε εντοπίσει έξι τομείς όπου θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή στο μέλλον, εκτός, μεταξύ των οποίων οι διαρκεί έρευνε τη Επιτροπή για το Διεθνές Εμπόριο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το σκάνδαλο Cambridge Analytica, μετά ε, την πρώτη προσφυγή που ουσιαστικά έχει υποβληθεί στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια και πρέπει να πω ότι η κοινή μας πίεση έχει φέρει αποτελέσματα για το διορισμό της διαμεσολαβήτριας, του διαμεσολαβητή μάλλον για την ε, σπίτι ιδιωτικότητας. Ο κύριος Κιθ Κράτ ε, έλαβε τη θέση του Υφυπουργού στο State Department Οπότε γίνεται ο μόνιμος ομόλογος και συνομιλητής μας για τα θέματα της ε, ασπίδας ιδιωτικότητας. Το πρόβλημα λοιπόν αυτό, αυτή η τρεκυμία για την ασπίδα ιδιωτικότητας είναι πλέον πίσω μας. Θα πρέπει βεβαίως όλα αυτά να περάσουν και από τη Γερουσία, αλλά η κυβέρνηση έδωσε κάποια απάντηση. Έχουμε περάσει ως προθεσμία στην, τα τέλη Φεβρουαρίου για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης. Εγώ θα φροντίσω να συναντήσω τον διαμεσολαβητή, τον κύριο Κετσό, το δυνατόν συντομότερα και αυτό γιατί θέλω να τον γνωρίσω, να δω τι άνθρωπος είναι και να το επιβεβαιώσω πόσο σημαντική είναι η δουλειά του για μας. Η έκθεση καταλήγει ότι η ασπίδα ιδιωτικότητα ε, ανταποκρίνεται στα πρότυπα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων, που είναι τώρα υψηλότερη από ό,τι θα ήταν χωρί την ασπίδα. Εδώ καλύπτονται εταιρείε ε, και στοιχεία ακόμα και πολύ μικρές και ορίζονται κανόνες για τη μεταφορά των δεδομένων. Σκοπός είναι να αποσαφινιστεί το πλαίσιο και η σχετική προσπάθεια θα συνεχιστεί. Οι συζητήσεις της ΕΙΠΑ για το Ομοσπονδιακό Σύστημα Προστασίας συνεχίζονται και θα συμμετέχουμε και εκεί. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε και άλλα βήματα για να ενισχύσουμε τα συστήματά μας με ισχυρά οριζόντια δικαιώματα και ανεξάρτητη διασυνοριακή ε, συμμόρφωση με τον νόμο, επιβολή του νόμου. Έχουμε συνονιθεί με τις ΙΠΑ για το θέμα αυτό και έχουμε αποστείλει και επιστολές για να συμμετάσχουμε στις δημόσιες διαβουλεύσεις τους. Ελπίζουμε να συνεχίσετε και εσείς τις συζητήσεις με τους ομολόγους και συνεργάτες στην Αμερικανική Γερουσία. Επίσης να στραφώ και στην Ιαπωνία να πω ότι η συμφωνία αντιστοιχία συγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα τεθεί σε... και τέθηκε ήδη σε ισχύ στις 23 Ιανουαρίου όπως και η απόφαση αμοιβές αναγνώρισης από την Ιαπωνία. Έτσι, με τη συμφωνία αυτή δημιουργήσαμε το μεγαλύτερο χώρο στον κόσμο για την προστασία των δεδομένων και την ασφαλή ροή τους. Αυτό έρχεται στην κατάλληλη στιγμή για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιαπωνίας. 1η ε, Φεβρουαρίου την Παρασκευή αυτή τη εβδομάδα συγκεκριμένα. Η φεβρουαριου την παρασκευη αυτη τη βδομάδα συγκεκριμενα η ιαπωνια με την απόφαση της ε, για τον πλήρη σεβασμό για τα προσωπικά δικαιώματα και την προστασία τους και φροντίζει για τη διάδοση των υψηλών ευρωπαϊκών προτύπων της προστασίας δεδομένων σε όλο τον πλανήτη. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο συμμερίζεται τη σημασία της απόφασης αυτής που δείχνει ότι όλα όλα τα βήματα που γίνονται για την προστασία των δεδομένων είναι σημαντικά. Η Ιαπωνία μετά από το GDPR για την ε, γενική προστασία των δεδομένων, το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων, είναι η πρώτη τέτοια περίπτωση. Και η προσέγγιση μα ήταν συνετή και ε, λελογισμένη για να φροντίσουμε η προστασία των δεδομένων να μην επηρεαστούν από το πώ εξελίσσονται οι διαβουλεύσει και οι διαπραγματεύσει για τα εμπορικά θέματα. Χρειάστηκε λοιπόν να γεφυρώσουμε κάποιες διαφορές απόψεων μεταξύ μας για την προστασία των δεδομένων όπως και στον τομέα, εμπορικό τομέα. Η Ιαπωνία όμως ε, έκανε αυτό που έπρεπε με τους συμπληρωματικού κανόνες όπως ονομάστηκαν και στα εμπορικά ζητήματα και στην προστασία των δεδομένων, δημιουργώντας μια ειδική δομή για τους Ευρωπαίους πολίτες ώστε να υπάρχει ε, επαρκής απόδοση δικαιοσύνης εφόσον χρειαστεί τα κατάλληλα ενδικά μέσα. Ως προς το ψήφισμα για το σχέδιο αποφασής μας και τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας ε, για προς το Συμβούλιο της Προστασίας Δεδομένων φροντίσαμε να τις θέσουμε και στην Ιαπωνία και να λάβουμε απαντήσει για το σύστημά του, διορθώνοντα αναλόγω το σχέδιο απόφαση. Η τελική απόφαση έχει μεταβληθεί, ιδίω ω προ τη στενή παρακολούθηση τη υλοποίηση του συστήματο κανόνων στην Ιαπωνία, με περισσότερη σαφήνεια στο πεδίο τη απόφαση, την προστασία τη μεταφορά δεδομένων, τον κύκλο ζωή τη και το καθεξής. Επιπλέον ρήτρε προσθέθηκαν για τα πρόστιμα, τι ποινέ και άλλε κυρώσει που μπορεί να χρειαστούν στην Ιαπωνική νομοθεσία. Περισσότερο λεπτομερεί εξηγήσει και περισσότερα από όσα ουσιαστικά πρότεινε το ψηφισμά σα έλαβε υπόψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ε, κλασική μορφή. Πολλές χώρες από την Ασία ήδη συζητούν ή προσαρμόζουν την ε, νομοθεσία τους για την προστασία των δεδομένων χρησιμοποιώντας πρότυπο τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων, τον GDPR. Έχουμε γίνει πηγή έμπνευση για να κοιτάξουν να συγκλίνουν ε, ήδη από τώρα προς τους κανόνες μας. Έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα πρότυπο ε, πολλή δουλειά βέβαια μένει ακόμα μπροστά μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φροντίσει να είναι καλύτερη η, επιβολή των κανόνων προστασία δεδομένων. Αν δούμε τι έγινε με το σκάνδαλο της Cambridge Analytica και το Facebook, θα καταλάβουμε ότι οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη σοβαρότητα στο ε, πλαίσιο του προεκλογικής εκστρατείας. Ο κανονισμός GDPR θα πρέπει να ε, χρησιμοποιηθεί και για τα προσωπικά δεδομένα στην διαδικασία των εκλογών και τα πολιτικά κόμματα να σέβονται του σχετικού κανόνε του κανονισμού. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κοινέ απειλέ για τα κάτι μέλη, όμω οι αρχέ των κρατών μελών ακόμη δεν έχουν συνεργαστεί ούτε συντονιστεί ούτε ανταλλάσσουν βέλτιστε πρακτικέ και πληροφορίε. Αυτό είναι ο λόγο που δημιουργήσαμε ένα προεκλογικό δίκτυο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και καλούμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν του φορεί για την προστασία δεδομένων που έχουν για να δημιουργήσουν δίκτυα σε διακρατικό επίπεδο. Το... Η κυρία Ήρινεκ, που είναι ε, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού ε, Συμβουλίου για την ε, Προστασία των Δεδομένων, στι 20 στι 21 Ιανουαρίου φρόντισε να ενημερώσει σχετικά του εκπροσώπου των 100 μελών. Επίση, να σα πω ότι την περασμένη Παρασκευή το Κορεπέρ ενέκρινε την απόφαση για την τροποποίηση του ιστορικού καταστατικού των ευρωπαϊκών κομμάτων, προβλέποντα συγκεκριμένε κυρώσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τι περιπτώσει παραβιάσεων των κανόνων προστασία προσωπικών δεδομένων. Πραγματικά ανυπομονώ για την υλοποίηση αυτού του επιπλέον του συμπληρωματικού νομοθετήματο. Επίση, ω προ τι εκλογέ. Η διαφάνεια στι διαφημίσει ε, ε, είναι ένα θέμα που μα απασχόλησε και αυτό καλέσαμε τι πλατφόρμε πληροφορική των 100 μελών να συγκλίνουν με του κανόνε μα. Είδαμε ότι υπάρχει τάση η παραπληροφόρεση και αντιδημοκρατικέ διαδικασίε να παίρνουν διαστάσει στην προεκλογική εκστρατεία, ε, καλλιεργώντα τον φόβο και άλλα αρνητικά συναισθήματα θέλουμε να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι Ευρωπαίοι ψηφοφόροι να προστατευτούν όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα. Η προσέγγιση μα είναι ιδεολογικώ ουδέτερη, όμω προασπίζεται και προφυλάσσει πλήρω την ελευθερία του λόγου. Κυρίε και κύριοι, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει επιβολή των νόμων μα και να υπάρχει ε, ανεξάρτητη και αμερόληπτη έρευνα με δικαστές και εισαγγελείς που να ε, κάνουν αποτελεσματικά τη δουλειά της έχουμε προτείνει το πακέτο για τα αποδεκτικά στοιχεία με τις ε, διαδικασίες της δικαστικής αρρωγή να μην είναι ακόμα αρκετά επιταχυμένες ε, και στο ρυθμό της ψηφιακής εποχής. Χρειάζεται να βελτιωθούν ε, με τρόπο ικανοποιητικό και για σκοπούς των ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων. Είναι πολύ σημαντικό το ένταλμα ερεύνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ακόμη οι λειτουργοί δεν τα γνωρίζουν καλά και δεν ξέρουν πώς να τα χειριστούν. Θα πρέπει λοιπόν και οι διοικητικές μηχανές να αρχίσουν να συμμετέχουν. Με μεγάλη χαρά βλέπω ότι η κυρία Σίπελ εντόπισε για εκείνη την ανάγκη για ε, διαφανέστερη και επιταχυμένη πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία με ένα τυποποιημένο έγγραφο ε, εργασίας. Έχω καταλάβει ότι και πολλά, ε, πολλοί πρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και ενδιαφερόμενοι έχουν επισημάνει τις μέρημνές του σχετικά και στα μέλη του Κοινοβουλίου. Οι υπηρεσίες μου λοιπόν είναι στη διάθεσή σας για να μιλήσουμε τους συνεργάτες σας ώστε να αποσαφινιστεί και να βελτιωθεί η πρότασή σας. Έχουμε κάθε κοινό συμφέρον να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ευρωπαϊκό πλαίσιο με ε, πραγματικά στοιχεία προστασία για να βελτιώσουμε την ψηφιακή πραγματικότητα όσων λειτουργούν εκεί και για όλου όσοι παρέχουν υπηρεσίε. Όμω ε, το κατεπήγον τη πρόταση παραμένει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα πραγματικό πλαίσιο και καμία νομική βεβαιότητα για τους ερευνητέ, του ανακριτέ, του πολίτε και τι επιχειρήσει. Επιπλέον υπάρχει κίνδυνος ε, σύγκρουση συμφερόντων όταν οι εταιρείε μπορεί να βρεθούν σε θέση να πρέπει να ε, σεβαστούν την νομοθεσία μια χώρα αλλά παραβιάσουν του νόμου μια άλλη. Αυτό είναι κατεξοχήν ένα πρόβλημα για του ε, παροχέ υπηρεσιών που λειτουργούν ταυτόχρονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΣΥΠΑ. Ε, υπάρχει η πράξη για τον ΕΦΟΣ, το Cloud Act, ε, τον ΕΠΑ, που ήδη ισχύει από πέρσι. Ο κοινό μα στόχο είναι να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει προστασία των προσωπικών δεδομένων και στι δύο πλευρέ και δικονομικέ διασφαλίσει, ώστε να προστατεύονται παρκώ οι πολίτε με διμερεί συμφωνίε. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιβεβαιώσει την υπευθυνότητά τη και τι αρμοδιότητέ τη εδώ. Γι' αυτό σκοπεύω να προτείνω μια εντολή για μια σφαιρική συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα, ώστε να υπάρχει πρόσβαση στα αποδεικτικά στοιχεία. Μετά το τέλο των διαπραγματεύσεων, το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει πρέπει να εγκρίνει ούτω ή άλλω την ε, πρόταση αυτή τη συμφωνία. Η συμφωνία αυτή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει επιπλέον ε, διασφαλίσει για όσου θέλουν ε, να προχωρήσει το πακέτο των ηλεκτρονικών αποδεκτικών στοιχείων. Επίση, θα πρέπει να έχουμε περισσότερα εχέγγυα σε σχέση με όσα ήδη ισχύουν σε σχέση με τη συμφωνία της, της την συμφωνία ομπρέλα εδώ θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι γίνονται πλήρω σεβαστά τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και σε ατομικό επίπεδο. Δεν θέλουμε να περάσουμε από το παραθυράκι το cloud act στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε να κάνουμε κάτι ανάλογο. Μα ενδιαφέρει να προασπιστούμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Επιτρέψτε μου τώρα να στραφώ σε έναν άλλο σημαντικό τομέα των δραστηριοτήτων μα, την αποτελεσματική καταπολέμηση του ξεπλήματο βρώμικου χρήματο. Σε αυτό το πλαίσιο θέλω να πω λίγα λόγια για, για την πρόσφατη έκθεση τη Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή για τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Εθαγένειας και τις σχετικά εθνικά προγράμματα. Ε, έχουμε ήδη εκφράσει τι ανησυχίε μα για την ασφάλεια και το ξέπλυμα βράμικου χρήματο και του κανόνε που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για την Ευρώπη, διότι αν μια χώρα πουλάει την ηθαγένειά τη, πουλάει και την ευρωπαϊκή ηθαγένεια ταυτόχρονα. Την ξεπουλάει στην ουσία. Τα συστήματα αυτά γίνονται ε, ανοιχτέ πύλε για όσου έχουν ε, το μπαράγια να πληρώσουν. Άρα, ε, επειδή είναι δυσανάλογο το θέμα αυτό να είναι απλώ εθνική αρμοδιότητα, η πώληση της ηθαγένειας θα πρέπει να απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο. Η έκθεση χαρτογραφεί τις ε, υπάρχουσες πρακτικές και εντοπίζει τους ενεχόμενους κινδύνους, όπως τις απειλές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως ό,τι αφορά την ασφάλεια, την, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά. Θα πρέπει να μην υπάρχει κανένας αδύναμος κρίκος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και να μην μπορεί ο καθένα να επιλέξει την υπηκέστερη δικαιοδοσία ή σύστημα. Ξέρουμε πώ ε, παρέχονται οι θεωρήσει και τα διαβητήρια. Ε, θα χρειαστεί όμω περισσότερη συνεργασία μεταξύ των μελών στην ανταλλαγή πληροφοριών για την ε, εξέταση των αιτήσεων όσων ζητούν διαβατήριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά στην περίπτωση που η πρώτη αίτησή του έχει απειριθεί. Θα πρέπει επίση να μην τα αφήσουμε αυτά ω αποκλειστικό προνόμιο των κρατών μελών. Θα πρέπει να γίνει ένα χρυσό κανόνα όποιο παίρνει την ευρωπαϊκή υπηκότητα θα πρέπει να έχει αυθεντική, πραγματική και ουσιαστική, ουσιαστικό δεσμό με τη χώρα όπου πήρε το διαπατηριό τη. Ελπίζω ότι αυτό ε, το βήμα θα γίνει ένα ε, κάτι που θα ξυπνήσει τα κράτη-μέλη, θα τα βγάλει από το λίθαργο για να αναλάβουν δράση ένα καμπανάκι που θα ε, ξυπνήσει τα κρατη Θα πρέπει να συνεργαστούν ε, οι εθνικοί εμπειρογνώμονες για το ε, για, τις συστηματικές, για τους συστηματικούς ελέγχους υγείας, για να γίνονται check-up δηλαδή και για τη σωστή ε, εφαρμογή των κανόνων. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξει πώς οι εθνικοί κανόνες είναι συμβατοί με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και να αναλάβει δράση εκεί που χρειάζεται. Αυτό είναι ένα από τα προσφατότερα παραδείγματα των ε, πρωτοβουλειών μας για να γίνει η Ευρώπη ασφαλέστερη, να δυσκολέψουμε τη ζωή των εγκληματιών και να καλύψουμε τα υπάρχοντα κενά. Ε, θέλουμε να επικαιροποιήσουμε του κανόνε μα για την καταπολέμηση του ξεπλήματο βρώμικου χρήματο και να του ενισχύσουμε. Θέλουμε επίση να ενισχύσουμε την εποπτεία της, ε, του ξεπλήματο βρώμικου χρήματο από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και έχουμε δημιουργήσει και την αρχή τη Ευρωπαϊκή Δημόσια Εισαγγελία. Ε, Βλέπω μάλιστα ότι προοδεύει σημαντικά η θέσπιση του οργάνου αυτού και το συζητήσατε μόλις νωρίτερα σήμερα. Επίσης, έχουμε ήδη διορίσει τον προσωρινό διευθυντή, ο οποίος θα φροντίσει ε, να γίνει σωστά η διαδικασία επιλογής των επιψηφίων για τον επικεφαλής της ε, Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ε, νομίζω ότι έχετε λάβει και την γραπτή επισκόπηση για το θέμα αυτό και από τον Κλοντ έμαθα μόλις τώρα ότι η Επιτροπή σας έχει ασχοληθεί εγκαίρως με το όλο θέμα της επιλογής του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο στόχο μα λοιπόν είναι η απόφαση αυτή να ληφθεί εντό αυτή τη θητεία. Τώρα για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο. Ζητήσαμε να προχωρήσει γρηγορότερα η υλοποίηση τη βασική νομοθεσία, βλέποντα τα πρόσφατα γεγονότα στην Γερμανία αλλά και άλλα παράπονα από άλλα κρατημέλη. Θέλουμε να υπάρξει πλήρη μεταφορά των σχετικών κανόνων και ενίσχυση τη εθνική νομοθεσία. Ελπίζω ότι θα υπάρξει θετική ανταπόκριση από την πίεση που ασκήσαμε. Σα ευχαριστώ επίση για την υποστήριξή σα το θέμα της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ε, μυστικών υπηρεσιών δίωξης οικονομικού εγκλήματος και τις δικές μας αρχές. Θέλουμε να υπάρξει αποτελεσματικότερη συνεργασία και σε αυτόν τον τομέα. Τέλος, να σας ενημερώσω για την αυτόνομη αξιολόγησή μας για τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου. Ξέρετε ότι οι επιτροπέ Πάνα και Τάξ 3 έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Ω χώρε προτεραιότητα θα έχουμε καταρτήσει κατάλογο μάλλον για χώρε πρώτη προτεραιότητα από τα τέλη τη περασμένη χρονιά. Χώρε ε, με τι οποίε έχει ασχοληθεί η ομάδα κατά τη του οικονομικού εγκλήματο και επίση και αυτόνομη αποτίμηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντα υπόψη τα πρότυπα της οδηγίας για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, καθώς και της μόνης ιδιοκτησίας. Εδώ με την ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό έχουν, έχουμε ήδη σημειώσει πρόοδο και τις επόμενες μέρες θα έχετε ε, περισσότερα νέα. Εδώ έκλεισα τις παρατηρήσεις μου και είμαστε διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ, Κλοντ. Ευχαριστώ. Επίτροπε, αναφερθήκατε προηγουμένω στην Ιθαγένεια και γι' αυτό θέλω να μιλήσω. Ε, Όπω και θέλουν να τα πουλήσουν τα μεγάλα λόμπι, δεν έχουν καμία σχέση, δεν έχει καμία σχέση το θέμα αυτό με τι επενδύσει. Εγώ προέρχομαι από τη Μάλτα, λέει η κυρία Μέτσολα, και ήμουν πάντα υπέρ των καλόπιστων ε, επενδύσεων, αλλά η, η πώληση ε, διαβατηρίων δεν είναι επένδυση. Ε, πουλάμε δηλαδή ένα διαβατήριο για, σε ανθρώπου που δεν έχουν καμία σχέση με τον λόγο, με λόγο χώρα, με πολύ σημαντικού ε, κινδύνους ε, διαφθοράς. Ε, δεν χρειάζεται μάλιστα καν να έχει κάποιος κάποια σχέση. Το άλλο μεγάλο ε, σημείο ε, πώληση είναι αυτό του κύριου Πρωθυπουργού, του κύριου Μουσκάτη. τη ε, Μάλτα, που πάει που ανά τον κόσμο λέει ότι το πρόγραμμά του είναι το μόνο το οποίο έχει την επίσημη έγκριση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το λέει αυτό, έτσι. Άλλο η θαγένεια, άλλο οι θεωρήσει και, και για τι παραμονέ. Διότι η θαγένεια είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αφαιρέσει κανείς. Μια φορά πληρώνεις και μετά εσύ και όλοι οι απόγονοί σου έχουν την ηθαγένεια σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό δηλαδή που αγοράζει κάποιος δεν, αγοράζει απλά, δεν είναι απλά ένα διαβατήριο, αγοράζει το δικαίωμα, το αναφέρετο να είναι πολίτης και αυτός και τα παιδιά του. Ελεύθερη κυκλοφορία, ελεύθερη ε, κυκλοφορία χωρίς θεώρηση, ε, μπορούν να έχουν επιχειρήσεις, κανόνες ανταγωνισμού, ακόμα και κανόνες ε, περί ψηφοφορίας, συμμετοχή στι εκλογέ και όλα αυτά χωρί να έχει απτό καμία σχέση το άτομο αυτό με καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χιλιάδε διαβατήρια πολλούνται τη στιγμή που οι λαϊκιστές προσπαθούν να βυθίσουν την Ευρώπη στην κρίση ε, και λένε ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια χούφτα γυναικών και παιδιών προσφύγων στα, πλοία. Στα... Αυτό δείχνει όλη την υποκρισία του όλου θέματος. Κυρία Πίτρο, πρέπει να καταλάβατε ότι το, το, Τί η απέτηση ε, διαμονής δεν γίνεται σεβαστή και όλη αυτή η μυστικότητα που υπάρχει για το πόσα απολούνται και σε ποιους ε, είναι πολύ επικίνδυνη. Υπάρχει θέμα ασφάλειας, θέμα διαφθοράς, θέμα ξυλίματο χρήματος με βάση τα που είπατε. Μπορώ να σας πω εγώ, μπορώ να πω εγώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμφωνεί με την πόλη διαβατηρίων. Δεν την καλύπτει. Ε, λέτε ότι δεν μπορείτε να σταματήσετε από νομική πλευρά. Τουλάχιστον μπορείτε να μα πείτε ότι αυτό το σύστημα που χρησιμοποιεί η χώρα μου δεν έχει την έγκριση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Μπέρκη Σίπελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και την Επίτροπο που είναι εδώ. Ξεκινήσατε μιλώντα ε, για το Privacy Shield και τη δεύτερη αναθεώρηση. Γνωρίζετε ότι υπάρχει μια έκθεση ε, της ε, ε, Υπηρεσίας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ε, θέλω να αναφερθώ σε κάτι που είπατε στην εισαγωγή σας. Το ένα αφορά τον διαμεσολαβητή, τον Ombudsman. Είπατε ότι γνωρίζουμε μάλλον πλέον ότι υπάρχει ένας μόνιμος Ombudsman. Αυτό είναι καλό νέο. Ε, την έκθεση του, της, προσωπικών, δεδομένων εδώ λέγεται ότι ο δημοσιολαβητής εξακολουθεί να μην έχει αρκετές εξουσίες απέναντι στις αρμόδιες αρχές και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσει της Χάρτας Θεμελιών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να σχολιάσετε σχετικά. Επίσης υπάρχουν κάποιοι κανόνες ε, για τις μεταφορέ, μεταφορές ε, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια έλλειψη υποχρέωσης οι οργανώσεις να ε, επιδεικνύουν τα συμβόλαια που ε, συνάπτουν με εταίρους από τρίτες χώρες για να μπορούμε να αξιολογήσουμε κατά πόσο αυτά τα συμβόλαια έχουν τις απαραίτητες κλίσεις ασφαλείας. Ε, θεωρείτε ότι υπάρχοντες κανόνες σχετικά με αυτά τα εμβάσματα ε, ε συνάδουν με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και κάτι ακόμα για το Privacy Shield Αναφερθήκατε στην FTC, η οποία δεν μπόρεσε να δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαραίτητες πληροφορίες ε, σχετικά με τις έρευνες για, το, για την Cambridge Analytica και το Facebook, ότι οι έρευνες συνεχίζονται. Μετά από κάποιους μήνες, σε έχετε λάβει πλέον κάποια νέα στοιχεία, κάποια περαιτέρω στοιχεία για την υπόθεση αυτή. Και κάτι άλλο. Αναφερθήκατε στο e-evidence. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, διότι ακόμα εξετάζουμε το επόμενο έγγραφο εργασίας. Το βασικό πρόβλημα που έχουμε, εγώ και κάποιοι συνάδελφοι τουλάχιστον, είναι ότι στο Ευρωπαϊκό Έντελμα Έρευνας μιλάμε για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πληροφορίες με κάποιους περιορισμούς, με κάποιε δικλείδε ασφαλεία. Όμω αυτοί οι περιορισμοί και δικλείδε ασφαλεία δεν βρίσκονται πουθενά στη νέα πρόταση. Έχοντα λοιπόν κατά νου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να συζητήσει και για συμφωνίες και για το Cloud Act, ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι με τέτοιου κανονισμούς, με τέτοιε συμφωνίε δεν θα νερώσουμε τα ζητήματα προστασία δεδομένων και τη δικλής ασφαλείας ό,τι αφορά την επιβολή του νόμου. Ε, εμείς θα εργαστούμε από αυτού, αλλά μένουν πολλά ακόμα ζητήματα που μένουν να εξεταστούν. Ευχαριστώ Μπίρκιτ. Μπίρκι, η, η Ναταλή Γκρίσμπεκ έχει το λόγο κανονικά, αλλά πρέπει να φύγετε, πρέπει να πάτε κάπου ε, πηγή. Η Ναταλή σε πειράζει να πάρει το λόγο η Άννα Γκόμες πριν. Σύντομα όμως. Ναι. Εκτός μικροφώνου η Γκόμες. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε και Επίτροπε. Συμφωνώ με τις ανησυχίες που εξέφρασε η συνάδελφος από τη Μάλτα και εκτιμώ ιδιαίτερα την έκθεση αυτή. Η περιγραφή του προβλήματος είναι πολύ καλή, όμως η έκθεση είναι αδύναμη στα συμπεράσματα, στις συστάσεις, στις δράσεις δηλαδή. Και, και με σοκάρει το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια σύσταση για την ανάγκη τα κράτη-μέλη ε, να προσέχουν τι γίνεται με τους ανθρώπους που έχουν, που έχουν διεθνείς κυρώσεις. Αυτό είναι πραγματικά εξοργιστικό. Όπως έχουμε ένα σύστημα όπως στη δική μου χώρα, στην Πορτογαλία, όπου εγώ ως Ευρωβουλευτής και οποιοδήποτε άλλος δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Σας ζητώ λοιπόν στις δράσεις σας αυτό που έχετε κατά νου, ζητείτε, ζητείτε δέουσα επιμέλεια από την Πορτογαλία. Θα μελετήσετε κατά πόσο υπάρχουν άτομα που υπόκειται σε κυρώσει στου καταλόγου αυτού, να μην πούμε και για άλλου εγκληματίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήσασταν και σύντομοι και ευχαριστώ Ναταλή που ήσουν καλή και άφησε την, τον, τη θέση σου. Ευχαριστώ Επίτρο, κυρία Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε. Ενδεχομένω μπορεί να μην ακούω, απαντήσω, να ακούσω τι απαντήσει, αλλά θα είναι εδώ η συνάδελφή μου, η βοηθή μου. Δύο-τρία πράγματα εν συντομία, διότι με τη Σοφή μοιράσαμε κάπως τα ερωτήματα από την ομάδα μας. Χθες γιορτάσαμε την Διεθνή ημέρα προστασίας δεδομένων στον Ευρωπαϊκό χώρο. Πάντα υπάρχει κάτι να γιορτάσουμε. Χθες όμως η χθεσινή ημέρα ήταν σημαντική σημαντικός εορτασμός για τους Ευρωπαίους πολίτες αλλά και για σας και για την Επίτροπο και για τις εργασίες της Επιτροπής μας. Οκτώ μήνες αφότου ξεκίνησε η εφαρμογή του περίφημου RGPD ε, που τελικά ε, γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτόν και πρέπει να συνεχίσουμε ε, να εξηγούμε, να εφαρμόζουμε ε, τις θεμελιώδεις ελευθερίες που προκύπτουν Περίπου 100.000 ε, προσφυγές έχουν γίνει έως τώρα προς τις αρχές προστασίας δεδομένων. Μόλις ε, τρεις έχουν, ε, οδήγησαν μάλλον σε κυρώσεις. Θέλω να ένα σχόλιο από αυτού, κυρία Επίτροπε, για το θέμα αυτό. Ποια είναι τα διδάγματα έως τώρα, λειτουργεί τελικά αυτή η νομοθεσία κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα δεύτερο ερώτημα σύντομο, παλιό ερώτημα βέβαια. Ε, τον Ιούλιο του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής ε, της ε, ε, ίσης μεταχείρισης εκτός αγοράς εργασίας μεταξύ προσώπων χωρίς διάκριση λόγω πεπιθήσεων, ε, ηλικίας, θρησκευτικής προτίμησης, ε, σεξουαλικής προτίμησης, τα γνωρίζουμε. Αυτά είναι, η οδηγία κατά των διακρίσεων 11 χρόνια μετά. Δύο δηλαδή θητείες αργότερα το Συμβούλιο ακόμα δεν έχει θέση. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι το Συμβούλιο συχνά αδρανεί σε αυτά τα ζητήματα, αλλά εδώ ε, πραγματικά είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Το Συμβούλιο εξηγεί ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε ομοφωνία, εντάξει, αλλά για ένα τέτοιο κείμενο κανονικά θα έπρεπε να επιτευχθεί. Εσείς και η Επίτροπε σκοπεύετε να κάνετε κάτι, γιατί και αυτό είναι κάτι που μιλάει στους Ευρωπαίους πολίτες, που δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, όπως και εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Αναφερθήκατε τώρα ότι θα αρχίσει να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ επανέρχομαι σε αυτό που λέω πάντα. Μας πήρε πολύ χρόνο να θεσπίσουμε αυτήν την εισαγγελία και βεβαίως ε, πρόκειται για ένα απαραίτητο εργαλείο για την καταπολέμηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας. Θα ήθελα να ξέρω, αφού του άκουσα τη Ρουμανική Προεδρία την περασμένη ε, εβδομάδα στην Επιτροπή Ελευθεριών, εάν συμμερίζεστε την ε, επιθυμία της Προεδρίας να υπάρξει επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκή Αγγελία και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας που είναι βεβαίω μια σύγχρονη απειλή αλλά είναι και μια απειλή που εξορισμού διασυνοριακή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Νάταλη. Κύριε Μπόνι. First of all, thank you very much. Uh, Καταρχάς ε, να σας ευχαριστήσω κυρία Επίτροπε για το συνεργασία που έχουμε στον τομέα των δικαιωμάτων και των αξιών. Ε, είχαμε και τον πρώτο τριμερή διάλογο. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία αυτή. Ε, αναφέρομαι κυρίως στο Συμβούλιο, αλλά πάντως με εσάς έχουμε σίγουρα μια πολύ καλή συνεργασία. Θέλω να τονίσω ότι ε, το, το επίτευγμα στον τομέα της ασπίδας ιδιωτικότητας είναι τεράστιο πραγματικά. Το συζητήσαμε και πριν από ένα χρόνο, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις και σας ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας σε αυτές. Επίσης, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι έπειτα από δικές μας πιέσεις το Υπουργείο Εμπορίου ξεκίνησε τη διαδικασία πιστοποίησης, αναδιοργάνωσης του πλαισίου και της διενέργειας, ξεκίνησε και τη διενέργεια κάποιων ελέγχων ε, επιτόπιων. Όλα αυτά είναι πολλά υποσχόμενα και πολύ θετικά δείγματα, αλλά βεβαίως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να επαγρυπνούμε και να συνεχίζουμε να πιέζουμε γιατί Τώρα, με την, ε, τώρα ε, θα περάσουν πολλοί μήνες μέχρι να ληφθεί η ε, οριστική απόφαση από την Γερουσία. Επίσης, θέλω να υποστηρίξω πλήρως με τη συνάδελφό μου την κυρία Μετσόλα και να συμφωνήσω μαζί της ότι θα πρέπει να υπάρχουν πολύ σοβαρότεροι και αυστηρότεροι κανόνες. Διαφανείς κανόνες. Είναι και απέτηση των πολιτών μας. Τέλος, για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Νομίζω ότι πρέπει η δουλειά αυτή να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό. Χρειάζεται να βρούμε τις σωστές λύσεις, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να αποφύγουμε μια ενδεχόμενη προσπάθεια να ξεκινήσουν διμερεί διαπραγματεύσει. Ευχαριστώ. Σόφι Ιντβελτ, um, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για όλα τα θέματα στα οποία αναφερθήκατε. Ερωτήσεις και παρατηρήσεις έχω να κάνω. Πρώτον, για το Privacy Shield. Προφανώς ε, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι επιτέλους θα υπάρχει ένας μόνιμος διαμεσολαβητής. Αν δείτε όμως τον ε, επιλεγέντα, αναφερθήκατε ότι θα είναι Φυπουργός περιβάλλοντος, ε, εμπορίου, ε, κυβερνήσεις ε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανοικοδόμης έχει και μια, δέκα άλλες ιδιότητες ο άνθρωπος αυτός θα τον ορίσει ο Τραμπ λοιπόν για να πάρει αυτές τις δέκα αρμοδιότητες πρώτον πόσο ανεξάρτητος θα είναι ο άνθρωπος αυτός και δεύτερον πόσο χρόνο θα έχουμε για να κάνουμε σοβαρή δουλειά και δεδομένου ότι πρόκειται και για πρώην επιχειρηματία, ε, δεν είμαι και πολύ βέβαιη τι είδους ε, εχέγγυα και διαπιστευτήρια έχει αυτός ο άνθρωπος για να είναι ο καταλληλότερος για αυτή τη θέση. Ε, να το πω ευγενικά, δεν έχω πιστεί. Δεύτερον, για την εντολή για την σύναψη συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης είπα, δεν θα σας ε, ε, κουράσω τώρα με τις δικές μου προσωπικές απόψεις. Θεωρώ πάντως ότι είναι πολύ κακή ιδέα, γιατί αυτό που ε, στην ουσία είναι το ζητούμενο είναι η κατάργηση του, των έμλατς, της, ε, της δικαστικής προσφυγής. Ε, ξέρετε, οι, οι σύντομες επιταχυμένες διαδικασίες είναι ίδιον των δικτατοριών. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Εμεί βέβαια πρέπει να δούμε την εντολή. Φυσικά η Κομισιόν θα πει «Ε, δεν, δεν μπορώ να σα δώσω την, τη στρατηγική. Μα η στρατηγική είναι άλλο πράγμα από την εντολή. Η, η εντολή είναι η δική σα πρόταση προ του Ευρωπαίου πολίτε. Δηλαδή τι θα διαπραγματευτείτε εκ μέρου των Ευρωπαίων πολιτών. Έχουν δικαίωμα να ξέρουν. Η εντολή δεν ταυτίζεται με τη στρατηγική. Οι Ευρωπαίοι πολίτε έχουν δικαίωμα να ξέρουν τι θα πάτε να διαπραγματευτείτε στο όνομά του. Δεύτερον, να μας ενημερώσετε για την σύμβαση της Βουδαπέστης που έγινε, η τελευταία ε, ενημέρωση σχετική έγινε πριν από τέσσερα χρόνια γιατί ξέρουμε ότι παρασκηνιακά συνεχίζονται κάποιες συζητήσεις για την αναθεώρηση της ε, σύμβασης ε, της Βουδαπέστης προκειμένου, ο απότερος στόχος είναι δηλαδή, να καταργηθούν τα έμλατ. Γίνεται λοιπόν μια διατλαντική προσπάθεια για την κατάργηση των ΕΜΛΑΤ. Νομίζω ότι είναι τελείω λάθο. Χρυσέ βίζε. Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπαν η Άννα και η Ρομπέρτα και εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει απαγόρευση των, χρήσεων, των χρυσών θεωρήσεων ή των χρυσών διαβαρτηρίων. Δεν είναι δυνατόν η ηθαγένεια να είναι εμπόρευμα προσπόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ μέχρι πρότινος έλεγα ότι χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια. Ε, δεν αρκεί. Α μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Πρόκειται για ένα κόκκινο χαλί που στρώνουμε σε εγκληματίε για να έρθουν εδώ και να γίνουν Ευρωπαίοι πολίτε. Εξηγήστε μου, γιατί κάποιο Ρώσος, και εγώ δεν μιλάω τώρα για μπάμπουσκες και τα λοιπά και τα ούτε για ρούβλια που είναι... Ε, ε, κρυμμένα σε παλιέ κάλτσες. Υπάρχει Ρώσος που, ήθελε, που είχε όνειρο τη ζωής του να γίνει μαλτέζο. Συγγνώμη, υπάρχουν άνθρωποι που πάνε στη Μάλτα και ζητάνε διαβατήρια. Το ίδιο και ενώ στι κάτω χώρε στις έχει έρθει ένας, ένας ε, εσείς γιατί πιστεύετε ότι πάνε οι άνθρωποι αυτοί στη Μάλτα και δεν έρχονται στις κάτω χώρες. Ε, μα συγγνώμη, άμα δίνεται ευρωπαϊκή ηθαγένεια, είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα ασφάλεια, είναι πρόβλημα επιβολή του νόμου, είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν, είναι πάντοτε πάρα πολύ αυστηρή όταν μιλάμε για επιβολή του νόμου. Ε, βγάλτε και το σωστό συμπέρασμα ότι δεν γίνεται αλλιώ. Η μόνη λύση είναι να απαγορευτούν οι πωλήσει διαβατηρίων τη ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Ε, Α δείξετε και επιτέλου λίγο θάρρο. Όχι απλά να λέτε μήπω θα μπορούσαμε να να, να προτείνουμε ή να παροτρύνουμε τα κράτη-μέλη σε αυτοσυγκράτηση. Όχι. Πρέπει να απαγορευτούν. Και πρέπει να απαγορευτούν για να προστατευτεί το κράτο δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από δυόμιση χρόνια, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ως δημοσιονομική αρχή, υιοθέτησαν προπολογισμό, ο οποίος συμπεριλέλαβε πρόταση για ένα ταμείο για την για την επίλυση διαφορών. Εδώ και δύο χρόνια σας κυνηγάω για να γίνει επιτέλους λειτουργική μια τέτοια αρχή. Επιτέλους φαίνεται ότι θα λάβουμε αυτή την πρόταση. Αλλά άμα το δείτε το, το κείμενο, ε, αλλά ξέρετε αυτά τα κείμενα πολλές φορές τα καταπίνει ο εκτυπωτής, ελπίζω να το πάρουμε εν πάση περιπτώσει, ε, το κείμενο αυτό ε, στην ουσία θα εξαντλείται στο να δοθούν κάποια χρήματα σε ΜΚΟ κοιό κτλ. Όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν μιλάω γι' αυτό. Ξαναλέω, τι ακριβώς έχουν αποφασίσει οι αρχές, οι δημοσιονομικές, είναι η θέσπιση ενός ταμείου για την επίλυση διαφορών, όπου πολίτες επιχειρήσεις και μη κυβερνητικέ οργανώσει θα μπορούν να προσφέρουν στα δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών του. Και ξέρω ότι η Κομισιόν υποστηρίζει αυτή την προοπτική. Γι' αυτό και περιμένω το συντομότερο δυνατόν να μα υποβάλλετε επιτέλου αυτή την πρότασή σα, οι υπηρεσίε σα, για να δούμε τι ακριβώ έχετε κάνει σε σχέση με αυτό που έχουν αποφασίσει οι συνομοθέτε, η Δημοσιονομική Αρχή. Και μια τελευταία παρατήρηση. Μιλήσατε για fake news και τα λοιπά και τα λοιπά, για ξένους πράκτορες που επεμβαίνουν και επηρεάζουν εκλογικά αποτελέσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμερίζομαι απόλυτα, κυρία Επίτροπε, τις ανησυχίες σας, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι πολλά από τα σκουπίδια, δηλαδή fake news, τα διαδίδουν όχι ξένοι φορείς, αλλά και ευρωπαϊκοί φορείς, όπως για παράδειγμα η Ουγγρική κυβέρνηση, η οποία ε, τα τελευταία και παρά τους κανόνες, τα τελευταία πέντε χρόνια η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή δεν έχει σηκώσει ούτε το δαχτυλάκι της για να κάνει κάτι για τα ψέματα που λέει ο Όρμπαν στους πολίτες του και στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψέματα που οδήγησαν μέχρι και στο Brexit. Επιτέλους σας γίνει μια πραγματική συζήτηση και επιτέλους αναλάβετε δράση για να τους αντιμετωπίσετε αυτούς. Μην έχετε στραμμένο το βλέμμα σας μόνο σε ξένους πράκτορες και φορείς που προσπαθούν τάχα να επέμβουν σε ευρωπαϊκές εκλογές. Γίνεται και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Επιτέλους, αντιμετωπίστε τα ψέματα που λέγονται και διαδίδονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Είπε κάποια πράγματα που και εμένα μου αρέσανε και θα μπορούσα να τα έχω πει και εγώ, Σόφη. Ευχαριστώ. Κάτι από αυτά που είπες ήταν η εντολή για διαπραγματεύσει με τη ΣΥΠΑ για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις. Ε, επίτροπε, θα μπορούσατε να μας πείτε εάν θα μπορεί το Κοινοβούλιο να ρίξει μια ματιά στο πώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις βάσει του κανόνα για τα απόρριτα έγγραφα και την ε, ε, δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά. Όχι, όχι, έχω κι άλλα. Συνάδελφοι, ξέρω ότι η Σόφη βγήκε από το ρεύμα του χρόνου της, αλλά δεν ήθελα να την κόψω. Συνάδελφοι, έχει κανένα ε, άλλο ε, διάθεση να παρέμβει και μετά θα δώσω το λόγο στην Επίτροπο. Σοράγια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Εγώ έχω μια τελείω διαφορετική ε, ερώτηση για την οδηγία της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Ντάλματος Ερεύνης. Από το 2011 ήμουν εισηγήτρια για την υλοποίηση ακριβώς της οδηγίας αυτής. Αυτό που αντιμετωπίσαμε ήταν ότι κανείς δεν γνώριζε η υλοποίηση μπορούσε να γίνει μέχρι το 2015. Και από 180.000 ε, διαταγές εντολές μάλλον μόνο μία ευρωπαϊκή ε, εκδόθηκε. Κανεί δεν τα ήξερε από τους υπευθύνου φορείς. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε αν ένα χρόνο μετά, εάν έχετε λάβει τίποτα μέτρα ώστε να ξέρουμε τι γίνεται με την προστασία των θυμάτων. Υπάρχει κάποιος που ασχολείται με την προστασία τους, οι αρχές που εργάζονται για τα θέματα αυτά. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καταρτήσει ένα σύστημα τρόου ή αρχείου για να μπορέσει να συλλέγει τα σχετικά στοιχεία από τα κράτη-μέλη και επίσης θέλαμε να ξέρουμε αν παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πώς προχωράει η υλοποίηση της οδηγίας και αν έχει ξεκινήσει παραβάση για δικασία των 100 μελών που την παραβίασαν. γίνεται καμιά προσπάθεια και από την κοινωνία των πολιτών για την οποία να έχει γνώση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώ υλοποιούν την οδηγία τα κατημέλη. Θα μπορούσα να συνεχίσω, αλλά επειδή δεν έχουμε χρόνο, νομίζω ότι πραγματικά υπάρχουν πολλά κενά εδώ. Για το πώ θα μπορούσε να χρησιμοποιείται αυτό το εργαλείο και την ανάγκη να το χρησιμοποιήσουμε και πλήρω. Ευχαριστώ πολύ, Σωράγια. Σε ευχαριστώ που ήσουν σύντομη. Είχε πολύ ζουμί όμω η ερώτησή σου. Να πω ότι μας μένει ο Χουάν Φερνάντο, η Λίδια, ο Γιουκά, ο κύριος Ζάντεφ, ο κύριος Γιουρέκ. Και μετά ολοκληρώνω. Ξέρω ότι όλοι μπορείτε να είστε ευσύνοπτοι, οπότε Χουάν Φερνάντο. Ναι, πολύ σύντομα. Βεβαίω μπορώ να είμαι τάχιστο, Επίτροπε Γιούροβα. Διότι η ερώτησή μου ουσιαστικά ταυτίζεται με κάποια από τα πράγματα που ήδη υπόθηκαν για την ασπίδα της ιδιωτικότητας ξεκίνησε η συζήτηση από την προηγούμενη θητεία του Ευρωκοινοβουλίου, ήμουν εδώ και θυμάμαι ότι ήδη από τότε προϋπόθεση για την επαναδιαγμάτευση μετά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ήταν ακριβώς η ετοιμότητα που θα έδειχνε η τότε κυβέρνηση Ομπάμα να δώσει κάποια απάντηση στι ευρωπαϊκέ ανησυχίε, στι ευρωπαϊκέ μέρημνε. Ιδίω αυτέ που εξέφρασε το Ευρωκοινοβούλιο γραπτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πώ έχουν διαμορφωθεί εδώ μεταξύ προοπτικέ, ήθελα να μου πείτε ε, εάν από τη συστηματική σας ανάλυση και αξιολόγηση ε, του πώς λειτουργεί η ασπίδη εάν μιλάμε για υποβάθμιση της αρχικής ατμόσφαιρας εντός της οποίας είχε συμφωνηθεί η πρώτη ασπίδα ιδιωτικότητας ε, με την προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ. Μήπως η αλλαγή της κυβέρνησης εκεί ε, εξηγεί την ε, δυσκολία και τη δυσφορία των μελών του Κοινοβουλίου που τα έχουν ήδη εντοπίσει και το γεγονός ότι ο διορισμός του διαμεσολαβητής της ΕΠΑ είναι μια προσπάθεια για να ε, υλοποιηθεί καλύτερα η ασπίδα προστασία από την Αμερικανική πλευρά, αλλά μπορεί να μην είναι αρκετή. Ευχαριστούμε, Χων Φερνάντο, που ήσουν τόσο σύντομο, Λίβια. Ευχαριστώ και μπράβο σας για τις μας δεσμεύσεις σα, για τα περισσότερα ντοσιέ που μα αναφέρατε και για το πόσο δύσκολη δουλειά έχετε φέρει σπέρα. Δεν μπορώ παρά να σας πω και εγώ ότι τα συζητήσαμε στο ΕΛΚ, το συζήτησε και η κυρία, το ανέφερε και η κυρία Μετσόλα. Εσείς προωθήσατε τον το αυτό και για το Facebook και, το Cambridge Analytica, και την Cambridge Analytica, το σχετικό σκάνδαλο. Τα, οι ψηφοφόροι λίγο πριν τις εκλογές ρωτούν για το θέμα αυτό και ρωτούν και για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο κτλ. Η δουλειά σας τέλος πάντων είναι πραγματικά ε, τη σημασία, για εμά και για τους ψηφοφόρου. Οπότε, εγώ σε αυτή την επιτροπή ασχολούμαι με το όλο θέμα των Ρωμά. Ε, μας ενδιαφέρει η ενδιάμεση αξιολόγησή σας και από όλες τις ε, πολιτικές ομάδες σκοπεύουμε να υποβάλουμε και ένα ψηφίσμα για την επόμενη Ολομέλεια. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι χρειάζονται περισσότερα αποτελέσματα από τις πολιτικές που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως τα κονδύλια που εκτελώνται. Η Ρουμανική Προεδρία κάτι πρέπει να κάνει και η Φινλανδική Προεδρία θα έπρεπε να αναλάβει μια γενικότερη πρωτοβουλία για τη φτώχεια. Στην Κροατική ΔΕ θα θέλαμε να ασχοληθούμε με τους φτωχούς των ε, Βαλκανίων διότι πιστεύουμε ότι η προσχώρηση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων εφόσον γίνει θα φέρει ένα τεράστιο σοκ σε χώρες που ακόμη δεν έχουν προτιμάσει τους πολίτες τους. Είναι πολύ φτωχοί οι άνθρωποι εκεί σε σχέση με τους περισσότερους στη Δυτική Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν κάτι να γίνει. Δεν θεωρείτε ότι κάτι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούσε να, να λάβει δράση γοργά ή είναι τελείω μη ρεαλιστικά αυτά που έχουμε σκεφτεί. Θα μπορούσαμε πυρημανικέ πρεδρέ να ελπίζουμε σε πρόοδο. Να μιλήσουμε για τα προγράμματα τη ανεργία, για την εκπαίδευση, για περισσότερη χρηματοδότηση, για πράγματα που θα μπορούσαν να προχωρήσουν καλύτερα. Υπάρχει λοιπόν περιθώριο του ερχόμενου 9 μήνε μέχρι τον Νοέμβριο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι θερμά συγχαρητήρια από μένα. Ευχαριστούμε και τελευταία είδη συνάδελφοι, ο κύριος Ζάντεφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Γιούροβα, έχω ένα ερώτημα για την οδηγία πρόσβαση στις πληροφορίες για τις περιπτώσεις ξεπλήματος χρήματος και άλλα εγκλήματα για τα οποία ζήτημα είμαι εισηγητής. Ένα από τα πιο αφιλεγόμενα σημεία της πρότασης είναι η εισαγωγή προθεσμιών για την ανταλλαγή πληροφοριών. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες και πολλές έχουν να κάνουν με τις διεθνείς πρακτικές. Δεν υπάρχουν διεθνή πρότυπα για προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών. Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τώρα ε, μονάδων <laughs> οικονομικού εγκλήματος. Ε, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έχει σκεφτεί να κάνει κάτι σε διεθνές επίπεδο για να δημιουργηθούν πρότυπα για την ανταλλαγή πληροφοριών. Λαμβάνουν χώρα διαπραγματεύσει στην ομάδα του ΕΓΜΟΝ για να υπάρξουν προθεσμίες εντός των οποίων θα πρέπει να ανταλλάσσονται αυτές τις πληροφορίες. Εγώ νομίζω ότι η εισαγωγή τέτοιων παγκόσμιων προτύπων θα ήταν επωφελής για τη διεθνή συνεργασία. Εάν λάβουμε υπόψη μας ότι το ξέφλυμα χρήματος, η, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας δεν έχουν σύνορα. Τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αισθήματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ παρακαλώ ο κύριος Τσίτσιρεκ. Ο κύριος Γιούρεκ. Ευχαριστώ πρόεδρε θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ζήτημα για το οποίο έχω μιλήσει και στο παρελθόν στην Ολομέλεια μπορεί να μην συζητήθηκε εδώ αλλά νομίζω πως ε, έχει τη σημασία του πολλές φορές τα κράτη-μέλη της Ένωσης έχουν ενθαρρυνθεί να επικυρώσουν τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, της Ισταμπούλ μάλιστα ε, δεχτήκαμε επιθέσεις γι' αυτό επειδή δεν τις επικυρώνουμε, η χώρα μας, ε, ε, ενώ δεν μπορούμε να εγκρίνουμε μια διεθνή συμφωνία που αντιβαίνει τις διατάξεις του συντάγματός μας. Το λέει αυτό το ε, βουλγαρικό συνταγματικό δικαστήριο. Αυτό αφορά και άλλες χώρες που, είναι, που βρίσκονται υποπίεση πάλι, θες, πάλι συνταγματικά ζητήματα προβάλλονται. Υπάρχουν λοιπόν όλες αυτές οι χώρες οι οποίε βρίσκονται υπό πίεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κανονικά η Κομισιόν συντονίζει. Δεν πιέζει έστω και εμέσω. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν σέβεται το κράτο δικαίου, δεν σέβεται επαρκώ τι μειονότητε και δεν υπάρχει αλληλεγγύη σε ό,τι αφορά τι ε, διμερεί σχέσει. Φτάνουμε στο τέλο τη θητεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποτέ δεν είναι αργά όμω για να διορθώσει κάποιο τα λάθο, τη λάθη του. Σα ενθαρρύνω λοιπόν, κυρία Επίτροπε, να κάνετε κάτι γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ όλου για την υπομονή σα. Είχαμε καθυστερήσει, είχαμε διακοπέ. Κυρία Επίτροπε, παρακαλώ, στο μέτρο του δυνατού, προσπαθήστε να απαντήσετε ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω στα ερωτήματα. Βέβαια, σε κάθε μία από τι ερωτήσει αυτέ ε, χρήζει μεγάλη συζήτηση πολύ σημαντικά θέματα και δύσκολα θα ξεκινήσω με αυτό που ρώτησε εσύ Κλοντ για την εντολή διαπραγμάτευσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω ότι τέθηκε και ένα ερώτημα σχετικό από την κυρία Ιντεβελτ είμαι βέβαιη ότι ενημερώσουμε έγκαιρα, θα ενημερώσουμε έγκαιρα ε, το Κοινοβούλιο. Αύριο θα εγκρίνουμε την εντολή, όχι την, την ερχόμενη εβδομάδα, στις 6 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε με βάση το, τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ ε, Κοινοβουλίου και Κομισιόν. Θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία που προβλέπεται, εν πάση περιπτώσει. Το Κοινοβούλιο θα ενημερωθεί άμεσα και πλήρω σε όλε τι φάσει διαπραγμάτευση, ε, όπω συμβαίνει στη σύναψη διεθνών συμφωνιών. Θα σα ενημερώσουμε λοιπόν μόλι ε, εκδοθεί η εντολή. Αυτή νομίζω είναι η διαδικασία. Θα σεβαστούμε πλήρω. ε, τα ε, τις απαιτήσει ε, διαφάνειας που υπάρχουν. Αυτό έχει να κάνει και με την δημόσια επικοινωνία μας. Είναι κάτι που αφορά τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν θέλουμε λοιπόν εδώ να παρθούν αποφάσεις ή να προχωρήσουμε ε, στο παρασκήνιο. Είναι γνωστή η διαδικασία που προβλέπετε και θα την σεβαστούμε. Λοιπόν, για το Privacy Shield ε, κυρία Σίπελ πρώτα είναι, είναι για τα γενέθλια σήμερα χρόνια πολλά είναι ένα θέμα πάνω στο οποίο πρέπει να εργαστούμε περαιτέρω στην αρχή είχαμε αυτή την, την προσφορά από τους Αμερικανούς για τη δημιουργία αυτού του Ινστιτούτου ε, ότι θα είναι κάποιος ε, ένα άτομο εμπιστοσύνη αυτό που θα θα υπόκειται στο Υπουργείο Εξωτερικών αλλά θα είναι ανεξάρτητος από την ε, ε, κυβέρνηση, την μυστικές υπηρεσίες, ε, αλλά και από τη μονάδα εντός της οποίας δημιουργήθηκε. Και έχουμε συμφωνήσει για μια διαδικασία που θα εγγυάται ότι οι προσφυγές Ευρωπαίων πολιτών θα εξετάζονται γρήγορα και δίκαια. Θα λαμβάνουν μια απάντηση σύντομα για το κατά πόσο τα δικαιώματά τους ε, έχουν παραβιαστεί. Ο δημοσιογραφητής ως τώρα έχει 31 προσφυγές πρέπει να έχει την απαραίτητη, απαραίτητη προσόντα ο δημοσιολαβητής το είχα πει την προηγούμενη φορά για μένα αυτός ο μικρός αριθμός προσφυγών δείχνει ότι δεν γνωρίζουν, δεν γνωρίζει ο κόσμος ότι μπορεί να προσφύγει. Δεν γνωρίζει ε, για ενδεχόμενες υποθέσεις παραβίασης των δικαιωμάτων τους. Ε, εάν υπάρχει κάποιο κενό λοιπόν είναι, έχει να κάνει με την ενημέρωση των πολιτών ότι υπάρχει δηλαδή αυτή η διαδικασία ότι υπάρχει αυτή η οδός που δημιουργήθηκε για, την, ε, ε, για να μπορούν να προσφύγουν και μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν ε, με εμπιστοσύνη. Τώρα, ε, έρχομαι τώρα πάλι στο θέμα του διαμεσολαβητή. Κατά πόσο ο κύριος Κρέτς θα μπορέσει να κάνει αυτή τη δουλειά του ε, πλήρως αυτό. Ελπίζω, ναι, θα έχει πολλά καθήκοντα. Ως τώρα υπήρξε μία προσφυγή δεν νομίζω λοιπόν ότι θα έχει και πολλά να αντιμετωπίσει. Εμείς περιμένουμε να κάνει σωστά τη δουλειά του. Είναι πολύ σημαντικό και να μπορεί να την κάνει και να την κάνει σε ένα πνεύμα εμπιστοσύνης. Θα πρέπει να περάσει βεβαίως και από τη Γερουσία. Ε, δεν θέλω εγώ να κρίνω να προδικάσω ότι δεν θα λειτουργήσει αυτή η ιστορία. Εμείς θέλουμε και αναμένουμε να λειτουργήσει. Τώρα για την ερώτηση της κυρίας ε, Σίπελ για, τις, ε, για τα εμβάσματα. Νομίζω ότι η απόφασή μας ξεκαθαρίζει και τα δύο ζητήματα αυτά. Και το θέμα των εμβασμάτων. Πάντα, πάντα ζητούμε ε, να υπάρχει συνένεση. Παρότι ε, Εάν ακόμα δεν χρησιμοποιείται μια διαφορετική διαδικασία που αφορά τρίτη χώρα. Χρειάζεται συνένεση. Εάν δεν υπάρχει συνένεση, δεν πρόκειται να υπάρχει μεταφορά. Περαιτέρω μεταφορά, όχι έμβασμα, περαιτέρω μεταφορά. Ε, κάθε φορά λοιπόν, ακόμα αν και η Ιαπωνία έχει μια συμφωνία με μια τρίτη χώρα, αυτό δεν αρκεί για μας. Έχουμε δηλαδή ενσωματώσει το σύστημα υποχρεωτική συνένεση για αυτές τις υποθέσεις. Τώρα πάντα θα ερώτημα της κυρία Σίπελ, το EFTC και οι έρευνες. Οι έρευνες είναι εν εξελίξη. Ε, με ρωτάνε συχνά γι' αυτό, για την Cambridge Analytica Η εταιρεία, από όσο ξέρω, δεν υπάρχει πια. Η συμμετοχή της πάντως στο Privacy Shield έχει ανασταλεί και το Facebook βρίσκεται υπό έρευνα. Ένα από τα ζητήματα, ένας από τους παράγοντες που εξετάζονται είναι το θέμα του timeline, του χρονολογίου. Διότι από όσο ξέρουμε αυτό έγινε στα πλαίσια του ασφαλού λιμένα και ουσιαστικά είναι η παραβίαση της νομοθεσίας της Αμερικανικής 2011 περί ιδιωτικής ζωής ε, αυτή που ισχύει εδώ η συμμετοχή λοιπόν του Facebook με βάση το Privacy Shield δεν πρέπει να επηρεαστεί από αυτό αλλά δεν μπορώ να προδικάσω τίποτα, η έρευνα είναι εξελίξη η FTC ξέρει πολύ καλά ότι ήμασταν υπόμονοι θέλουμε να γνωρίζουμε την αλήθεια για το τι συνέβη γιατί είναι κάτι που επηρέασε, αυτό είναι βέβαιο πια, εκατομμύρια Ευρωπαίους. Πάλι για το Privacy Shield, ο κύριος Μπόνι, α δεν είναι εδώ ο κύριος Μπόνι, συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουν προς τα Αμερικανοί, είναι και η απάντηση του κύριο Λόπες Αγγιλάρ, Βεβαίως, η αλλαγή στην Αμερικανική κυβέρνηση είναι ο λόγος για τον οποίο εγώ προσωπικά ανησυχώ. Ήδη ήταν δύσκολα με την κυβέρνηση Ομπάμα να φτάσουμε σε συμφωνία για αυστηρούς κανόνες, ε, για μια έτσι ενεργητική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την προστασία των ε, ε προσωπικών δεδομένων στο αμερικάνικο έδαφος στην αρχή υπήρχε μια τάση να υποτιμήσουμε ε, το Privacy Shield ως ένα σύστημα που θα εγγυόταν τα προσωπικά δεδομένα από αμερικανικής πλευράς ε, και σε μεγάλο βαθμό αυτό έχει να κάνει με την προσέγγιση σε ό,τι αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής αυτή καθ' αυτής καθ' αυτής. Ξέρετε ότι στην Αμερική είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όμως ε, αλλάζουν οι καιροί, όπως είπε και ο Μπομπ Ντίλαν η περίπτωση νομίζω της Cambridge Analytica είναι αυτή που άνοιξε μια νέα δημόσια συζήτηση αντιδράσεις υπήρξαν και στο Κογκρέσο και και νομίζω ότι σύντομα θα υπάρξει κάποια νομοθεσία που θα μοιάζει με το GDPR με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων, θα είναι ένα ομοσπονδιακό νόμο καινούριο. Τώρα κύριε Λόπε Αγγιλάρα έχετε δίκιο. Εμεί θα είμαστε ικανοποιημένοι μόνο με δύο προποθέσει. Είτε θα υπάρξει ένα GDPR ε, σε αμερικάνικο στυλ, αυτό είναι κάπως αγαθό όμως για την ώρα. Εμείς αυτό ζητάμε, ομοσπονδιακή νομοθεσία που να είναι ισοδύναμη με το GDPR αυτό επιζητούμε εμείς, γι' αυτό στείλαμε και σχόλια ε, στη διαδικασία διαβούλευση στη δική τους και βεβαίως από εκεί πέρα θα ήταν ικανοποιητικό επίσης αν είχαμε πρόσβαση σε πληροφορίες στις μυστικές υπηρεσίες τους, στις διάφορες ε, στους διάφορους άλλους οργανισμού πώ ε, έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και πώς τα επεξεργάζονται. Αλλά δεν έχουμε τέτοια πρόσβαση πρέπει να βασιστούμε ε, στη δική τους νομοθεσία, στο πώς την εφαρμόζουν αυτοί, ε, στην αρχή του ενδεχόμενου κόστους, ε, που είναι κάτι αντίστοιχο με την αρχή αναλογικότητας και επικορικότητας τη δική μας. Και να πω κάτι ακόμα, δεν έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και σε ευρωπαϊκό έδαφος. οπότε δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες ούτε στις ΗΠΑ. Γι' αυτό η λειτουργία του δημοσιολαβητή εδώ, αυτού του θεσμού, είναι κρίσιμη. Βασιζόμαστε ε, σε αυτή τη νέα, σε αυτό το νέο θεσμό, σε αυτό το πρόσωπο. Θα είναι ο άνθρωπος που στις πολιτείες θα έχει πρόσβαση στις πληροφορίες τις οποίες θα χρειαζόμαστε εμείς. Είναι περίπλοκο το σύστημα, αλλά νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει όλε τι δυνατότητε έτσι ώστε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερε πληροφορίε ε, και να υπάρχουν και εργαλεία ε, και από την Αμερικανική πλευρά. Ο κ. Λόπε Αγκιντάρ, κ. Μπόνι, οι Αμερικανοί πρέπει να κάνουν περισσότερα. Ναι, εμεί του πιέζουμε να είναι πιο ενεργοί στο θέμα αυτό. Έχουμε και αυτή τη νέα διαδικασία, κάποια τεχνολογία, για να αξιολογήσουμε τη συμμόρφωση των εταιριών με τους κανόνες του Privacy δεν είναι μια διαδικασία να εξελίξη. Δεν είναι μια απόφαση που πάρθηκε και τελείωσε. Και, τελείωσε. και βασιζόμαστε στους Αμερικανούς να κάνουν αυτά που πρέπει. Όχι. Ε, παρακολουθούμε, εποπτεύουμε, θα επανέλθουμε σε ένα χρόνο για να δώσουμε μια έκθεση, μια αναφορά ειλικρινή για το τι έχει συμβεί με την εφαρμογή. Υπό την κυβέρνηση του κ. Τραμπ πάντως ε, αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι θα είναι δύσκολο. Όταν ξεκινήσαμε τη δεύτερη ε, αναθεώρηση εδώ στις Βρυξέλλες είχαμε μια πολύ ισχυρή αμερικανική αντιπροσωπεία που εμφανίστηκε. Ήταν και ο Υπουργό Εμπορίου, ο διαμεσολαβητής, ε, ο επικεφαλής της FDC, πρέπει να πω ότι είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι από αυτήν την προσέγγιση που ακολουθούν. Τώρα για την ηθαγένεια. Ακούστε, ναι, οι διερμηνήσεις ενδεχομένω θα χρειαστεί να φύγουν σύντομα και θα πρέπει να συνεχίσουμε στα αγγλικά. Λυπάμαι γι' αυτό μόλις ενημερώθηκα σχετικά. Συνεχίζω στα αγγλικά, εσείς αγγλικά μιλάτε, ναι, βεβαίως. Όμως ε, οι δημιουργοί θα πρέπει σιγά σιγά να φεύγουν. Διαπιστώσετε, έχετε διαπιστώσει ότι έχουν βελτιθεί τα αγγλικά μου. Ναι, επειδή κάνετε παρέα μαζί μου, παρότι δεν λέω καλά το όνομά σου εδώ και πέντε χρόνια. Πολλά γίνονται εδώ μεταξύ μας και βεβαίως τα αγγλικά σας βελτιώνονται. Συγγνώμη, συγγνώμη, αυτό ήταν ε, ένα αστείο. Οι διερμήσεις σας αφήσουν δυστυχώς. Γεια σας από εμάς. Καλό βράδυ. The option of, of, of doing and writing. Uh, Roberta, I know you're keen for